Dear colleagues. Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Καθίστε. Πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να καλωσορίσω εδώ τον επαναδιορισμένο Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας, τον κύριο Δεγκίντος. Όπως ξέρετε, η συνάντηση αυτή είναι κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Ρέτζι και ΕΚΟΝ στα πλαίσια του διαφορετικού διαλόγου με την Επιτροπή βάσει του άρθρου 23 του κανονισμού για τα διευθυντικά ταμεία. Γνωρίζετε ότι ο διάλογος αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και οι συντονιστές αποφάσισαν και ενέκριναν την απόφαση στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου να έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τους Υπουργούς Οικονομικών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. και αυτό για την δράση που τους ζητήθηκε να αναλάβουν και επίσης για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο που θα έχει η ενδυνάμει αναστολή των βιβλίων των διαφορετικών ταμείων. Γι' αυτό διοργανώσαμε αυτή τη συνεδρίαση και να δώσω το λόγο στην φίλη και συνάδελφο πρόεδρο της Επιτροπής Ρέτζη για επιπλέον εισακτήριες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Γκουαλτιέρη. Καλησπέρα. Ε, καλημέρα σε όλους, δεν ξέρω τι να πω. Ε, είμαστε οι δύο αυτές οι επιτροπές στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να διοργανώσουμε την ακρόαση των Υπουργών Ισπανίας και Πορτογαλίας τους αξιότιμους κυρίους Ντεγκίντος και Σεντένου που περιμένουμε λίγο αργότερα. Να προσθέσω μετά τα λόγια του συναδέλφου ότι χρειαζόμαστε ημέν τους δε και συναντούμε τους υπουργούς σε κέρια στιγμή όταν ε, οι δύο χώρες έχουν υποβάλει τα σχέδια προπολογισμού τους ε, για το 2017, ένα μήνα περίπου μετά, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πρώτον και κατά δεύτερον, προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει πρόταση για αναστολή των διαθωτικών κονδυλίων ή και όχι για τα δύο αυτά κράτη-μέλη. Μετά συνεδρίαση και συνάντηση με του δύο επιτρόπους, αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Κατάινων, και την Επίτροπο Κρετσού που είναι υπεύθυνη για την περιφερειακή ανάπτυξη, θέλουμε να συνεχίσουμε. Και συνεχίζουμε τη δουλειά μας με την παρουσία των δύο υπουργών. Έχω τη χαρά τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεγκίδος, Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας. Υπουργέ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Δυστυχώς, ως συνήθως, δεν έχουμε χρόνο. 10 λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή. Ε, es siempre un honor comparecer ante las comisiones del Parlamento Europeo. Ήρθα εδώ ε, για, να για να αναφερθώ στα βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη σας στα πλαίσια του διαθρωμένου διαλόγου για την πρόταση σχετικά με τα διαθροτικά ταμεία και την ενδεχόμενη ε, κατάργησή τους για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στο ευρύτερο πλαίσιο της, των οικονομικών εξελίξεων και να αναφερθώ στη δέσμευση της χώρας μου έτσι ώστε να μπει τέλος ε, στο υπερβολικό ε, έλλειμμα. Η Ισπανία είναι από τις Χώρε που έχουν πληγεί σημαντικά από την οικονομική κρίση. Από το 2008 έω το 2013 το ΑΕΠ στην Ισπανία μειώθηκε κατά 9%. Καταστράφηκαν 3,5 εκατομμύρια θέσεις εργασία. Χάθηκαν. Ε, σε, ένα, σε μια διεθνή οικονομική συγκυρία εξαιρετικά εχθρική, η Ισπανία ξεκίνησε μια φιλόδοξη στρατηγική οικονομική πολιτική ε, εξυγίανση, εξυγίανσης, δημοσιονομικής εξυγίανσης και διαδροτικών αλλαγών. Έχουμε εξυγιάνει τον χρηματοοικονομικό τομέα, έγινε μια μεταρρύθμιση τη ε, ε, αγοράς εργασίας, πήραμε και μέτρα για να αυξηθεί ο ανταγωνισμό σε πολλού τομεί τη οικονομία. Αυτή την περίοδο αποδείξαμε ότι δεσμευόμαστε ε, με τις συστάσεις αναχώρα που μας έχουν απευθυνθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η Ισπανία είναι από τις χώρες της Ένωσης που τηρεί περισσότερο τις συστάσεις αυτές. Ήταν αποτελεσματική από τη στρατηγική. Το 2013 ξεκίνησε μια διαδικασία ανάκαμψης η οποία ενισχύθηκε τα δύο τελευταία χρόνια. Το ΑΕΠ ε, έχει τρία τρίμηνα συνεχόμενης αύξησης και σε δύο τρίμηνα πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε στο επίπεδο πριν την κρίση. Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας, η μεταρρύθμιση τη αγορά εργασία ήταν πολύ σημαντική. μπορούσαμε να δημιουργήσουμε θέσει εργασία ε, ευθύ εξ αρχή με την ανάκαμψη. Από την αρχή του 2014 έχουμε δημιουργήσει πάνω από 1,5 εκατομμύρια θέσει εργασία. Και η ανεργία έχει μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια ανθρώπου περίπου. Το 2015 ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό ό,τι αφορά τα οικονομικά επιτεύγματα και το 2016 συνεχίζεται η ίδια τάση. Το ΑΕΠ ε, αυξάνεται σε ρυθμούς πάνω από 3%, το διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Έτσι λοιπόν η Ισπανία μεταξύ των χωρών με τους μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης ε, μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών της Ένωσης. 600.000 θέσει εργασία έχουν, φτιαχτεί, έχουν δημιουργηθεί του τελευταίους μήνε και έχουν μειωθεί, 300, έχουμε μειωθεί κατά 300.000 η ανεργία. Ταυτόχρονα έχουμε μια πολύ σημαντική διόρθωση των, των μακροοικονομικών ε, στοιχείων. Η, ε, το ισοζύγιο πληρωμών είναι πλέον σε πλεόνασμα πάνω από 2% από ένα έλλειμμα που υπήρχε. Έχουμε επίσης πάνω από 10% αύξηση του ΑΕΠ. Η, ε, το χρέος έχει μειωθεί κατά 0,5% στον τομέα των οικοδομών, στις οικοδομήσεις αλλά και σε άλλους τομείς έχουμε μία ανάκαμψη και στον τομέα των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Επίσης υπάρχει μια βιωσιμότητα σε δημοσιονομικό επίπεδο. Η δημοσιονομική προσπάθεια που κάναμε ε, είναι αναμφισβήτητη. Το δημοσιονομικό έλλειμμα έφτασε στο 9,6% ε, και έχει μειωθεί στο μισά το 2015. Είμαστε μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης ε, μεγαλύτερης δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτή η σημαντική μείωση του ονομαστικού ε, έγινε σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης ε, περιορισμένη στην Ισπανία με αρνητικό πληθωρισμό και με μια οικονομική συγκυρία ε, εχθρική. Αυτό είχε επιπτώσεις ε, βεβαίως στο δημοσιονομικό έλλειμμα του 2015 0,5% σε σχέση με άλλες χώρες παρεμφερείς, με παρεμφερείς οικονομικές καταστάσεις ε, εξαιρετικές ε, ελήφθησαν υπόψη αυτέ τι εξαιρετικέ περιπτώσει. Έκανε μια σημαντική διαθροτική δημοσιονομική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια η Ισπανία. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η βελτίωση ήταν πάνω από 4% του ΑΕΠ στην περίοδο 2012-2015 και αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο έχουμε πάνω από 1% βελτίωση. Όμω, όπω λέει η ίδια η Κομισιόν, η διαθροτική προσπάθεια τη προσπάθεια τη Ισπανία υποτιμάται για λόγου μεθοδολογία του υπολογισμού η μεθοδολογία της, της Κομισιόν δεν λαμβάνει υπόψη της, τον αντίκτυπο, τον πραγματικό στις μεταρρυθμίσεις ε, των μεταρρυθμίσεων ε, στις, ε, στους ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν λαμβάνει υπόψη επίσης ε, ο πληθωρισμός. Ιδιαίτερα για χώρες όπου υπάρχει αποπληθωρισμός, όπως στην Ισπανία. Εάν λάβουμε υπόψη μας το κενό αυτό ονομαστικά, το output gap, η δημοσιονομική προσπάθεια θα ήταν του 5, του 5% του ΑΕΠ για την λόγο λόγω περίοδο. Αυτό σημαίνει μια προσπάθεια 1,25% το χρόνο, πολύ πάνω από τις απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ισπανία δεσμεύεται να σεβαστεί τους δημοσιονομικούς και οικονομικούς κανόνες της Ένωσης. Και αυτό φαίνεται και στην απάντηση της κυβέρνησης ε, στην, προσ... Ε, ε, προεδοποίηση του Συμβουλίου για να λάβουμε υπόψη μας την απόφαση προειδοποίησης του Συμβουλίου, η υπηρεσιακή κυβέρνηση ε, πήρε μέτρα για να εγγυηθούμε ότι θα πετύχουμε το στόχο για το έλλειμμα για το 2016. Σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο ε, περιφερειών έχουμε αλλάξει τον προπολογισμό ε, σε ό,τι αφορά το, την ε, πληρωμή σε δόσεις του των, του φόρου επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά άλλα, άλλα, άλλους φόρους που αφορούν ε, την κληρονομιά έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε και την φοροαποφυγή. Αυτά τα μέτρα αποφέρουν καρπού, όπω δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μα. Εκτιμούμε ότι οι δημοσιονομικέ επιπτώσει των μέτρων αυτών είναι πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2016. Πάνω από 1% δηλαδή του Ισπανικού ΑΕΠ, κάτι που θα μα επιτρέψει να πετύχουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για το 2016 ό,τι αφορά το, το έλλειμμα. 4,5% δηλαδή και να πετύχουμε και τον στόχο του ερχόμενου έτου που είναι 3,1%. Και κύριε όπω ξέρετε η αναστολή των διατροφικών τομείων η ενδεχόμενη μετά την απόφαση του ΕΚΟΦΗΝ του Ιουλίου ε, αυτή η απόφαση ε, ε έχει να κάνει με δύο διαδικασίε ε, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ένα ε, πρόστιμο. Στι 8 Αυγούστου το ΕΚΟΦΗΝ αποφάσισε να ακυρώσει το πρόστιμο για την Ισπανία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι για την ακύρωση του πρόστιμου και το Συμβούλιο και η Κομισιόν ανέφεραν τι πολύ σημαντικέ μεταρρυθμίσει που έκανε η Ισπανική κυβέρνηση από το 2012 σε, ένα, σε μια οικονομική συγκυρία δύσκολη και τι πολύ σημαντικέ δημοσιονομικέ προσπάθειε που έγιναν για να, για να διορθωθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα. Όλα αυτά ισχύουν και σήμερα και για τη διαδικασία που μα απασχολεί τώρα. Όπω λέει και ο κανονισμό των διευθυντικών ταμείων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των κρατών μελών, ιδιαίτερα το επίπεδο ανεργία. Παρά την καλή εξέλιξη τη αγορά εργασία στην Ισπανία, χρειαζόμαστε 1,5 εκατομμύρια θέσει εργασία ακόμα για να φτάσουμε στο επίπεδο απασχόληση που υπήρχε πριν αρχίσει η κρίση. Ε, η Κομισιόν λοιπόν ελπίζουμε να κάνει μια θετική αξιολόγηση τη δράση τη Ισπανία με βάση τα μέτρα που πήραμε ω κυβέρνηση. Τώρα με μια κυβέρνηση εκλεγμένη ε, εμείς δεσμευόμαστε εκ νέου να μπει τέλος ε, στο, υπερβολικό έλλειμμα ε, ως το 2018. Ε, σύντομα θα εγκρίνουμε ε, το δημοσιονομικό για το, τον προπολογισμό για το 2017, έτσι ώστε να φτάσουμε σε 3,1% δημοσιονομικό έλλειμμα το 2017 και να, έχουμε κάνει μια προσπάθεια 0,5% σε διαφορά του ρυθμού ανάπτυξη. Τα διαφορετικά ταμεία ε, και η αναστολή τους ε, δεν θα ισχύσει εφόσον παρθούν απαραίτητα, με, τα απαραίτητα αποτελεσματικά μέτρα. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Η Ισπανία λοιπόν είναι η χώρα που αναπτύσσεται περισσότερο από τις μεγάλες οικονομίες, το διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης έχει γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματο και ονομαστικά και διαθροτικά και εξακολουθούμε να δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τη δημοσιονομική προσπάθεια. Και αυτό το αποδεικνύει ότι ακόμα και η υπηρεσιακή κυβέρνηση πήρε μέτρα για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ισπανία είναι το πιο σαφέ παράδειγμα ότι μπορούμε να επανέλθουμε στην ανάκαμψη, στην οικονομική ανάπτυξη με εντό τη Ένωση χάρη στι μεταρρυθμίσει. Αυτή τη στιγμή μακροοικονομικά ε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε ό,τι αφορά στοιχεία τη Ισπανία και στο τραπεζικό επίπεδο δεν υπάρχουν ανησυχίε. Έτσι λοιπόν η αναστολή ε, των διαθροτικών ταμείων θα ήταν, δεν θα είχε νόημα και θα ήταν αντιπαραγωγικό. Θα στέλναμε ένα λάθο μήνυμα σε σχέση με αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Δεν θα λάβανε υπόψη τι βασικέ προτεραιότητε τη οικονομική πολιτική που αυτή τη στιγμή ε, ε, έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μια στιγμή όπου υπάρχουν κίνδυνοι, όπου υπάρχει αβεβαιότητα και για την οικονομία, την παγκόσμια, αλλά και για τι ευρωπαϊκέ χρηματαγορέ το να τιμωρηθεί η χώρα που έχει κάνει τις πιο, πιο, σημαντική, πιο σημαντική ανάκαμψη σε οικονομικό επίπεδο είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται και η Ευρωοικονομική, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη. Η πρόεδρο. σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα συνεχίσουμε τώρα προχωρώντας στον πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές της Επιτροπής Ρέτζι. Συζητήσαμε πώς να οργανώσουμε την ακρόαση και καταλήξαμε ότι θα ακούσουμε πρώτα τις ερωτήσεις των συντονιστών που δεν μπορούν να υπερβούν το 1,5 λεπτό ο καθένας και θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Βαν Νίστελ Ρόι που είναι ε, συντονιστής της ομάδας του Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια κύριε Υπουργέ για τον εκ νέου διορισμό σας στην Ισπανική κυβέρνηση. Συγχαρητήρια επίσης για την εξαιρετική περιφερειακή πολιτική που ε, εκτελείται ε, στην Ισπανία εδώ και χρόνια. Έχετε λάβει ε, βραβεία, το Regio Star, κατά επανάληψη. Και συγχαρητήρια επίσης και στη βάση των πληροφοριών που μας δώσατε και που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι εύκολη η δουλειά της Κομισιόν. είτε μηδέν αναστολή ή καθόλου αναστολή. Αυτή είναι βέβαια, η Κομισιόν είναι η αρμοδία για να κρίνει τα όσα είπατε. Την τελευταία φορά είπατε, είπατε στο τέλος δηλαδή, να μην ε, επιβάλλουμε τιμωρία στα λάθος πρόσωπα στους δικαιούχους των κοινωνικών προγραμμάτων. Αλλά εδώ έχω μια ερώτηση. Ο Επίτροπος είπε την τελευταία φορά ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις. Όμως, εάν αναστείλετε την εκτέλεση ενός προγράμματος, πόσο καιρό θα χρειαστείτε για να το ξαναρχίσετε. Είχαμε μία περίοδο που δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και οι χώρες έβαζαν τότε το χέρι στην τσέπη για να, βγάλουν το, να καταβάλουν τα υπόλοιπα. Αυτές είναι οι δυο ερωτήσεις. Πάντως ήδη αισθάνομαι πολύ καλύτερα από ό,τι στην τελευταία συνάντησή μας. Ευχαριστώ. Ο κ. Κοζολίνο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Έχει το λόγο. Είναι πραγματικά περίεργο να πρέπει να συζητήσουμε μέσα σε αυτό το μακροοικονομικό πλαίσιο που έχει παρουσιαστεί, διότι εδώ και δύο χρόνια υπάρχει η ενοποίηση. Τα δεδομένα είναι ιδιαίτερα θετικά και θα έπρεπε και ως προς την ε, νομοθεσία να μην χρειάζεται να ανοίξει καν η κουβέντα για την αναστολή της αποστολής των ε, κονδυλίων των διευθυντικών ταμείων. Παρ' όλα αυτά φτάσαμε και σε αυτό το σημείο και καταλαβαίνουμε πόσο δυσάρεστη είναι αυτή η συζήτηση, αυτή, αυτός ο διάλογος και η άποψη που έχει κυκλοφορήσει και έχει ακουστεί ήδη πολύ και στη συζήτησή μα με του επιτρόπου για την περίπτωση τη Ισπανία αλλά και τη Πορτογαλία, δεν υπάρχουν οι προποθέσει για την ε, αναστολή των ε, διευθυντικών κοντιλίων. Παρ' όλα αυτά, για σκοπού ε, καλή συζήτηση. Αρνητικό αντίκτυπο πρέπει να πω ότι θα έχει απλώ και μόνο η συζήτηση που κάνουμε για την ενδεχόμενη αναστολή των ειδικών κονδυλίων. Και θέλω εσεί να μου πείτε τι επιπτώσει θεωρείτε ότι είχε αυτή η θεωρητική συζήτηση που για μένα δεν έχει λόγο ύπαρξη. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχει καν η περίπτωση αναστολής για την Ισπανία. Ευχαριστώ, Λούερ της ομάδας ECR. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ ε, τον ε, κύριο Τεγκίντος που είναι παρόν σήμερα, η ομάδα μου των Ευρωπαίων ε, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών χαιρετίζει την ανάλυση της κυβερνήσεως από τον Μαριάνο Ραχώη και τους συνεργάτες του μετά από ένα έτος αβεβαιότητας. Υποστηρίζουμε την απόφαση να μην αναστέλουν οι πληρωμές <clears throat> των διαδοτικών ταμείων διότι θα προκληθεί επικίνδυνο προηγούμενο και ίσως να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που αναμένουμε, εφόσον θα επιβαρυνθούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί. Και στον διαθέσιμο χρόνο δεν έχουμε βέβαια τη δυνατότητα να επεκταθούμε. τελευταία, τα τελευταία νούμερα που έχουμε δείχνουν ότι η ισπανική ανεργία τον Ιούλιο του 2016 ήταν υψηλότερη και από αυτήν της Ελλάδος προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει από 6,4 δισεκατομμύρια σε 8,4 δισεκατομμύρια τις ενισχύσεις για τους νέους και επειδή η Ισπανία λαμβάνει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μπορείτε να μας δώσετε πληροφορίες σχετικά με κάποια προγράμματα που θεωρείτε ότι δεν αποδίδουν και ίσως μπορούν να καταργηθούν και να κατευθυνθούν τα ε, κονδύλια σε άλλα προγράμματα τα οποία να αποδίδουν. Ευχαριστώ. Άλντε Γιακόβτσιτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριοι Υπουργοί, επιτρέψτε μου να πω εξ ονόματος ε, της ομάδας μου, δηλαδή των φιλελευθέρων, πόσο ικανοποιημένοι είμαστε που βλέπουμε τις θετικές τάσεις να διαμορφώνονται καθαρά πλέον μετά από την κρίση που 2008 και που έπληξε τόσο βαριά τόσες πολλές χώρες. Μετά από τις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις, χαίρομαι που δύναμη να συμπεράνω ότι όντως αναφαίνονται ή διαφαίνονται θετικές τάσεις. Γνωρίζουμε καλά ότι η κρίση ε, χτύπησε τις χώρες της Μεσογείου και εγώ προερχόμαι από την περιοχή αυτή του κόσμου και γι' αυτό χαίρομαι που βλέπω τώρα θετικές τάσεις. Ρωτώ, πώς ακριβώς σχεδιάζετε να εφαρμόσετε τους κανόνες που σας επιβάλλουν να εφαρμόσετε. Κανόνες που εμείς έχουμε θεσπίσει οι ίδιοι βεβαίως. Με ποιον τρόπο θα το κάνετε και ποιες εγγύσεις μπορείτε να δώσετε για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα του ελλείμματος. Μιλήσατε για την μείωση του δημοσίου χρέους. Γνωρίζουμε ότι η χρήση κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής και των διαφορετικών Ταμείων συνολικότερα είναι απόλυτα αναγκαία και για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Αυτό είναι καθαρό. Θα θέλαμε ωστόσο να έχουμε κάποιες συγκεκριμένε εγγύησει για τους επόμενους μήνες και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας για το σχέδιο εφαρμογής των κανόνων που όπως είπα έχουμε θεσπίσει εμείς οι ίδιοι για τους εαυτούς μας. Ευχαριστώ. Από την ομάδα της Ενωμένης ΕΕ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η δική μας θέση, η θέση της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς είναι γνωστή. Είναι γνωστή σε όλους. Είμαστε κατά, ε, επί της αρχής ήδη, για την ε, μακροοικονομική αυτή εξέταση και έχουμε δώσει το σχετικό αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια τη τελευταία θητεία. Βεβαίω το γεγονό ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο σήμερα, σε αυτή την κατάσταση που είναι τελείω ε, ανευλογική, σημαίνει ότι λήφθησαν κάποιε αποφάσει στο μεταξύ. Υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει ευθύνη και στο επίπεδο του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, που υπό την ηγεσία τη δεξιά των σοσιαλιστών και του κέντρου καταλήξαμε να, καταλήξαν να αποδεκτούν αυτούς τους, αυτή την ε, μακροοικονομική ρεσιμότητα. Ε, ε, εδώ οι αποφάσεις του Συμβουλίου και της δικής σας κυβέρνησης έχουν ακριβώς το ίδιο μερίδιο στις ευθύνη όταν αυτή την ερεσιμότητα την πρότεινε το Συμβούλιο. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια ήταν η θέση της Ισπανικής κυβέρνησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αν αγωνιστήκατε κατά αυτής της ερεσιμότητας ή αν συμφωνήσατε είτε υποπίεση είτε λόγω των πεπιθήσεών σα. Επίσης θέλω να μου πείτε ποιε είναι οι δραστικές περικοπές τις οποίες αναγκαστήκατε να κάνετε για να υποκύψετε στις απαιτήσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Και ποιες είναι οι νέες προσπάθειες που προβλέπετε να επιβάλλετε στο λαό της Ισπανίας, ο οποίος έχει ήδη υποφέρει πολλά δεινά από αυτή την πολιτική λιτότητα. Και εν τέλει ήθελα να ξέρω εάν έχετε ε, αξιολογήσει τον αντίκτυπο μιας ενδεχόμενη αναστολής, την οποία θεωρούμε τελείως άκερη από πλευρά μας, μια ενδεχόμενη ε, αναστολής των κονδυλίων στις εξόχω απόκεντρε περιοχές. Ευχαριστούμε. Κυρία Βάνα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Υπουργέ που δεχθήκατε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς οι πράσινοι ε, θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να παίξει ενισχυμένο ρόλο στη συζήτηση αυτή. Και εμείς θεωρούμε ότι η απειλή αναστολή των πληρωμών των διαθετικών ταμείων θα οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα, διότι έτσι τιμωρούνται οι περιφέρειες. Και ιδίω οι περιφέρειες εκείνες που έχουν περισσότερο ανάγκη τις επενδύσεις για να ξεφύγουν από την κρίση. Για παράδειγμα, με πρόθεση της απασχόλησης. Ιδίω στην Ισπανία, είπατε και εσείς κύριε Υπουργέ, ότι ήδη έχετε λάβει αυστηρά μέτρα, ιδίω στο περιφερειακό επίπεδο, για να ικανοποιήσετε τους ε, κανόνε του συμφώνου. 80% των εξοικονομήσεων που έχουν γίνει έω τώρα έχουν γίνει στις περιφέρειες. Δηλαδή οι περιφέρειες έχουν φορτωθεί μέγα μέρος των περικοπών. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν οι μέχρι τώρα εξοικονομήσεις σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο. Πώς κατανεμήθηκαν, πώς κατανεμήθηκαν σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο και αν πρόκειται να κοπούν και άλλα κονδύλια τώρα, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη, στην φτώχεια, στην απασχόληση, και ιδίω για την επίτευξη των τόσο σημαντικών στόχων τη Ευρώπη 2020. Τελευταία ερώτηση. Σε ορισμένε χώρε βλέπουμε ότι τα ευρωπαϊκά διαθεωτικά ταμεία είναι οι τελευταίε επενδύσει που απομένουν πλέον και που γίνονται από το δημόσιο. Ισχύει αυτό και για την Ισπανία. Κατά τα λοιπά, θεωρώ, όπω και πολλοί που μίλησαν πριν από μένα, ότι το Συμβούλιο πρέπει να διακόψει αμέσως την ε, διαδικασία αυτή σε βάρος της Ισπανίας και Πορτογαλίας για να προστατεύσει τις περιφέρειες. Ευχαριστώ κύριε Ντεμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ που είστε εδώ. Η δική μου αντιπροσωπεία των πέντε αστέρων από την αρχή της θητείας έχει ε, με δρυμύτητα διταχθεί ε, στο Ευρωπαϊκό Εξάμενο και τους κανόνες του. Όμως, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου από την ίδια πολιτική Παράταξε με τον ε, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γιούνκερ, έχουν ουσιαστικά επιβάλει αυτή την πολιτική λιτότητα και τους ε, περιορισμούς ε, του προπολογισμού με μια φαντασιακή ουσιαστικά σταθεροποίηση της οικονομίας. Αυτό κινδυνεύει να έχει σοβαρότατο αντίκτυπο σε όλους τους συμπατριώτες των ιδίων των κυβερνώντων ακόμα. Εδώ λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχει κάνει συζήτηση για αυτή την ενδεχόμενη αναστολή. Ελπίζω, Υπουργέ, η δική σας κυβέρνηση να αλλάξει την δική της τάση σε σχέση με το παρελθόν. Και μία ερώτηση ε, για το άρθρο 23 εδάφιο 10. Λέγεται ότι πρέπει να υπάρξει ενισχυμένη πλειοψηφία για να ληφθεί η απόφαση εντός ενός μήνα από τη στιγμή της υποβολής της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρείτε ότι υπάρχουν οι για να συμβεί κάτι τέτοιο. Θεωρούμε ότι μια οριστική διέξοδο όπως όπω προβλέπεται από το άρθρο 23, εδάφιο 16, θα μπορούσε να είναι αυτή τη αναθεώρηση του άρθρου μετά την υποβολή έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω προβλέπεται για το 2017. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει νέα νομοθετική πρόταση. Δεν θέλουμε στη χώρα σα να επαναληφθεί το θέατρο παραλόγου, το οποίο ε, αναγκάστηκε να παίξει ο Ιταλό Πρωθυπουργό. Με διάλογο αδιέξοδο στην ε, πραγματικότητα με διαπραγματεύσεις χωρίς ουσία που πολλές φορές προκαλούν ε, τους μηδιασμούς αλλά τελικά καταλήγουν σε δραματικές εξελίξεις για, τα, για τους βασικούς χαρακτήρες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να, να φροντίσετε η αρμάτα, σας, η σας να μην ακολουθήσει την κατεύθυνση που έχει ήδη δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κύριο Γιούνκερ και τον, την ψευδολιτότητά του και να αλλάξετε τη στάση σας εδώ ήδη από τη συζήτηση ενώπιον του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει πρέπει η όλη κατάσταση να ξεκαθαριστεί. Διότι η Ισπανία και η Πορτογαλία εφαρμόζουν τα μέτρα που μόνο ακαδημαϊκοί έχουν προβλέψει, αλλά στην πράξη δεν δίνουν κανένα αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Μπριά, εκτός αν κάνω λάθος. Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα από τους συντονιστές της Επιτροπής Ρέτζιο. Θα ήθελα τώρα να σας ζητήσω κύριε Υπουργέ να απαντήσετε σε 8 λεπτά σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε και κύριοι ευρωβουλευτές. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω κάπως διότι πολλές ερωτήσεις έμοιαζαν. Κάποιες ανέφεραν ποιες ήταν οι επιπτώσεις της αναστολή των διαθροτικών ταμείων για την Ισπανία και την οικονομία της και κάποιες άλλες που έχουν να κάνουν με τους κανόνες και την, το σεβασμό των κανόνων αναφερθώ πρώτα σε αυτό το δεύτερο. Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικοί οι κανόνες. Τους κανόνες πρέπει να τους σεβόμαστε και να τους τηρούμε. Ιδιαίτερα εφόσον τους έχουμε αποφασίσει όλοι, όλοι μαζί. Η Ισπανική κυβέρνηση λοιπόν θεωρώ ότι τηρεί τους κανόνες. Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση που να έφερε σε πέρα μια τόσο σημαντική αλλαγή ε, στην οικονομική της συμπεριφορά στην Ευρωζώνη τα τελευταία πέντε χρόνια. Η Ισπανία πριν από πέντε χρόνια κατέστρεφε θέσεις εργασίας 700.000 το χρόνο. Είχε ξεκινήσει μια δεύτερη κρίση, το τραπεζικό της σύστημα δημιουργούσε φόβους, η χώρα δεν ήταν ανταγωνιστική και είχαμε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα πάνω από 9% του ΑΕΠ. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3%. Θα δημιουργηθούν 700.000 θέσεις εργασίας. Έχουμε ε, το, το πληρωμών το οποίο είναι πλεονασματικό. Το τραπεζικό μας σύστημα δημιουργεί πλέον καμία ανησυχία για την Ευρωζώνη και έχουμε διορθώσει όλες τις μακροοικονομικές ανισορροπίες μας. Έτσι λοιπόν αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δικασίας μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, εντατικής, ε, ονομαστικά το, μειώσαμε κατά 50% με συνεισφορά όλων των, των διοικήσεών μας ε, σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης και αυτό έγινε με έναν τρόπο που επέτρεψε να συνεχιστεί η οικονομικη ανάπτυξη. Επαναλαμβάνω εδώ και 13 τρίμηνα έχουμε ανάπτυξη. Είναι το πιο σαφές παράδειγμα του πώς μπορεί ε, μία χώρα σε κρίση να ανακάμψει χωρίς υποτίμηση να δημιουργήσει θέσει εργασία, να δημιουργήσει ανάπτυξη και να δείξει ότι σε μία νομισματική ένωση τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί μπορούν να λυθούν με την κατάλληλη οικονομική πολιτική. Έτσι λοιπόν Πέρα από το θέμα των κανόνων για την αναστολή ε, των διαθροτικών ταμείων και του προστήμου υπάρχει μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που είναι σημαντικό να την τονίσουμε. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή δεν προκαλεί καμία ανησυχία, καμία βεβαιότητα για τη μακροοικονομική οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης. Σε μια ε, λεπτή χρονική στιγμή, κρίσιμη σε μια στιγμή που υπάρχουν αβεβαιότητε, υπάρχουν ανησυχίε, υπάρχουν λαϊκισμοί παγκοσμίω. Η Ισπανία λοιπόν είναι ένα παράδειγμα του πώ μπορεί να αντιστραφεί μια τέτοια κατάσταση. Βεβαίω μένουν πολλά να γίνουν, το ξέρουμε. Έχουμε ε, ευάλωτα σημεία, βεβαίω. Έχουμε χρέο κοντά στο 100% του ΑΕΠ. Έχουμε ένα ποσοστό ανεργία τη τάξη του 19%. Ήταν 27 βέβαια, πριν από τρία χρόνια αλλά εξακολουθεί να είναι αυτή τη στιγμή λίγο κάτω από το 19%. Και βεβαίως η Ισπανία πάντα έδειξε τη δέσμευσή της απέναντι στους κανόνες. Μία και κυβέρνηση, όπως είπα προηγουμένως, μπόρεσε να πάρει μέτρα που οδήγησαν σε επιπλέον έσοδα για τον προπολογισμό της τάξης των 9 δισεκατομμυρίων κάναμε μεταρρύθμιση στο, σε ό,τι το των επιχειρήσεων και αυτό θα, θα μας φέρει πόρους που θα ξεπεράσουν ε, αυτά που προβλεπόταν. Oh, θα φτάσουμε στα 9 δις, ενώ είχαμε προβλέψει 8,3 δις. Ταυτόχρονα, μεταξύ των διαφόρων δημοσίων διοικήσεων, έχουμε μοιράσει το βάρος ε, των περικοπών και της μείωσης των δαπανών. Αυτό όμως που πραγματικά θα εγγυηθεί το μέλλον ε, και που θα εγγυηθεί το σεβασμό των δημοσιονομικών κανόνων είναι η διατήρηση των ρυθμών ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Και αυτό νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο έγινε σαφές ότι είναι εφικτό με βάση τις πολιτικές που ακολουθήσαμε. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Ναι, ε, εμείς βεβαίως ε, δεσμευόμαστε για, για τους κανόνες ακόμα και με του κανόνε που δεν συμφωνούμε. Αλλά είναι κανόνε όλων. Έτσι. Κάποιοι κανόνε μα αρέσουν και κάποιοι άλλοι δεν μα αρέσουν. Στην νομισματική ένωση όμω πρέπει κανεί να κάνει πολλέ προσπάθειε. Ε, υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Να προχωρήσουμε με την Τραπεζική Ένωση. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ταμείο ενιαίο για την εγγύηση των καταθέσεων. Πρέπει να έχουμε μέσα εργαλεία για να μειωθεί ο κίνδυνος, το ρίσκο. Αυτός είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις για το τι σημαίνει για την Ισπανία η αναστολή ε, των ε, διαδροτικών ταμείων. Μιλάμε για περίπου 1,2 δις αφορά πολλούς τομείς της οικονομίας πολλά σχέδια όπως ξέρετε είναι αντικείμενο χρηματοδότησης ε, των προπολογισμών του εθνικού προπολογισμού και των τοπικών προπολογισμών και μια τέτοια αναστολή πέρα από τον πραγματικά αχρίαστο στιγματισμό της Ισπανίας ε, θα είχε και αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Όμως πέρα από τις ε, επιπτώσεις αυτές επιτρέψτε μου να πω ότι το να επιβληθεί ένα πρόστιμο ή να ανασταλούν τα ταμεία ε, πραγματικά θα ήταν ένα χτύπημα ψυχολογικό για, για, για μας, για το λαό μας που, έχουν κάνει, που έχει κάνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια και που αρχίζει να βλέπει το φως το τέλος του τούνελ. Θα ήταν δηλαδή ένα λάθος μήνυμα, θα ήταν ε, μια μορφή όχι εξετελισμού αλλά πάση πτώση θα επηρέαζε σίγουρα το ηθικό ε, του πληθυσμού της Ισπανίας και τη Πορτογαλίας. Φαντάζομαι το ίδιο πρέπει να ισχύει. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τι τεράστιε προσπάθειε που έκανε η Ισπανική κοινωνία, τι τεράστιε προσπάθειε ε, για να ξεπεραστεί μια πολύ βαθιά κρίση, την πιο βαθιά κρίση τη ιστορία μα. Είπαμε προηγουμένω από την αρχή τη κρίση ω τα μέσα του 2013 χάσαμε 9 μονάδε του ΑΕΠ ε, χωρί προηγούμενο αυτή η κρίση και 3,5 εκατομμύρια θέσει εργασία και όταν καλύψαμε σχεδόν το σύνολο του ΑΕΠ, του, των ε, απολύων του ΑΕΠ και πάνω από το μισό των θέσεων απασχόλησης που χάθηκαν, τώρα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επιβάλλουν ένα πρόστιμο, κάτι που δεν έγινε τελικά, ή να αναστείλουν τα δευτερικά ταμεία είναι κάτι το οποίο ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Ελπίζω εσείς κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να ακούσατε τις ε, απαντήσεις. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη, τον συναδελφό μου. Ευχαριστώ. Πρώτος ο μιλητής μας από την Επιτροπή Οικονομικών, εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα είναι ο κύριος Σάλβα. Ευχαριστώ. Ε, είναι προφανές ότι η Ισπανία είναι μία από τις οικονομίες που έχει τις πιο υψηλούς δημούς ανάπτυξης. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η ανάπτυξη είναι στην καρδιά της πολιτικής της δράσης. Έτσι λοιπόν είναι προφανές και το είπαν πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές ότι η Ισπανία είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα σημείο αναφοράς. Η Ισπανία δηλαδή έκανε αυτό που, το αναλογούσε, αυτό που της αναλογούσε. Και βεβαίω είναι και θέμα αξιοπιστία τη Ευρώπη, των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα αξιόπιστε το να παγώσουμε τη χρηματοδότηση της Ισπανίας πραγματικά θα ήταν ένα πλήγμα για την εξοπιστία της Ένωσης και των θεσμών της και όπως ελέγχθη προηγουμένως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναθεώρηση του, της μεθοδολογίας υπολογισμού διότι δεν λήφθη υπόψη είναι ο αποπληθωρισμός. Ε, σας είδα αισιόδοξο κύριε Υπουργέ και εγώ συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας. Θα ήθελα μάλιστα να είμαι ακόμα πιο αισιόδοξο. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι είναι εφικτό να μειωθεί ακόμα περισσότερο το έλλειμμα κάτω από 4,6% φέτος και αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις ε, για τον υπολογισμό του ερχόμενου έτους. Ευχαριστώ. Σα Σας ευχαριστούμε πολύ, Περβάνς Μπερές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε. Στα πλαίσια του διαφορετικού διαλόγου, νομίζω, το Ευρωκοινοβούλιο ασχέτως του ότι ψηφίστηκε στην προηγούμενη θητεία, δείχνει εδώ την χρήσιμη συνεισφορά του για να επηρεάσει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην προχωρήσει, στις, ε, να μην προχωρήσει χωρίς καμία αναστολή στην ε, αναστολή των ε, κονδυλίων, των κονδυλίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζω να ακούσει και να τις ορθές προτάσεις που γίνονται εδώ σε αυτή τη συζήτηση και να περάσει στη μηδενική εφαρμογή. Όμως, από την παρουσίασή σας, αυτό που με εξέπληξε ήταν η μνήα στην ανάκαμψη στον κατασκευαστικό κλάδο στη χώρα σας. Ξέρουμε ότι είναι ένας κλάδος, ένας τομέας πολύ εκτεθειμένο, υπερεκτεθειμένο στην Ισπανία, με μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό. Ίσως διαφορετικά να ήταν χρήσιμο να μας πείτε λίγο περισσότερα για τις συνθήκες ανάκαμψης που έχετε διαδεί και την βιωσιμότητα που προβλέπετε. Επίσης, για την εξέλιξη της αγοράς εργασίας και τον κίνδυνο να υπάρχει εξέλιξη στην εργασία των μηδενικών ορών. Ευχαριστούμε. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές από την Επιτροπή ΕΚΟΝ έχουμε κάποιον, όχι από τους φιλελεύθερους. Καλό απόγευμα κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα καταρχήν να σας συγχαρώ ε, για την νέα θητεία σας. Ελπίζουμε αυτή να είναι ευτυχής και για τους Ευρωπαίους πολίτες και τους Ισπανούς. Θα αναφερθώ στη συνέχεια στο παράλογο της πρότασης αναστολής ε, των ταμείων, θα το πω και στην Πορτογαλία της προηγουμένως, στη συνέχεια μάλλον, αλλά επειδή ξέρω τα πράγματα από μέσα ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής ανησυχώ. Ανησυχώ και για την Ευρώπη και για την Ισπανία. Αναφερθήκατε βεβαίως ε, στα μακροοικονομικά στοιχεία τα οποία είναι θετικά ότι βεβαίω υπάρχει αυτή η βελτίωση, να αναγνωρίζουμε, αλλά το πρόβλημα που έχει η Ισπανία ήταν, είναι ένα πολύ μεγάλο διαφορετικό πρόβλημα, εξαιρετικά δίσκαμπτο και εξακολουθεί να λέει βεβαίως η ότι θα πετύχει του στόχου τη η Ευρώπη, αλλά δεν αντιμετωπίζει το πραγματικό πρόβλημα. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο δεν μπορούμε να το σταματήσουμε χωρίς μεταρρυθμίσει των, ε, των διοικήσεων, των εθνικών διοικήσεων, πάντα, πάντα θα, θα ε, υποσχόμαστε πράγματα που δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Ε, όπως ξέρετε, αυτή τη στιγμή ε, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα που πήραμε από το φόρο των επιχειρήσεων φέτος. Είναι <laughs> δηλαδή κάποια πράγματα που είναι μπαλώματα. Δεν θα λοιπόν να ξέρω ποιο είναι οψίες από αυτού, το διαφορετικό επίπεδο δηλαδή. Ευχαριστώ από την ΚΟΕ ο κύριος Διέγας. Δεν είναι εδώ. Παρακαλώ. Ναι, καλό σας απόγευμα. Παλώμα Λόπες πολύ θέατρο έτσι, σε αυτά τα ευρωπαϊκά φόρα. Απειλές, δεσμεύσεις, κάρτες που βγαίνουν. Λες και η κυβέρνησή σας κύριε Ντεγκίντος δεν συμμερίζεται το σχέδιο των Βρυξελών. Δηλαδή ιδιωτικοποίηση των συντάξεων, καταστροφή του δημόσιου τομέα, κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι τα ίδια κόμματα αυτά που υποστήριξαν και τις, ε, τα, τις συνθήκες ε, σταθερότητας. Ήσασταν υπέρ των μέτρων ε, για την οικονομική διακυβέρνηση και το κυρώσει στο 2011 και το 2012. Και η Ισπανία μπορεί να μείνει αυτή τη στιγμή χωρίς περιφερειακά και διαθροτικά ταμεία. Εσείς τιμωρείτε τους λαούς, όχι τις κυβερνήσεις. Διότι εσείς συμμερίζεστε τις πολιτικές αυτές. Αυτό το κοινοβούλιο έχει πει πολλές φορές ότι είναι κατά του παγώματος των ταμείων. Είναι πολύ απλό πείτε ότι δεν δέχεστε, δεν δέχεστε την, τον εκβιασμό των, των θεσμικών οργάνων. Δεν είπατε τίποτα κύριε Ντεγκίντος, από πού θα βγουν ε, τα 5,5 δισεκατομμύρια ε, περικοπών ε, που συζητήσατε στο κύριο Γκρουπ χθε από τις συντάξεις και τι θα κάνετε με τις λοιπές συντάξεις, μάλλον ε, προτάσεις θα συνδέεται με την απασχόληση, το Ταμείο Ενεργείας διότι οι θέσει που έχετε δημιουργήσει είναι ε, εύθραυστες, είναι προσωρινές. Δεν μίλησατε για την παραγωγικότητα. Η παραγωγικότητα από ό,τι πρόσθεσε στην κυβέρνηση μένει πολύ χαμηλά. Ε, υπάρχουν και οι τοπικές και επιφερειακές κοινότητες. Θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται ο νόμος Μοντόρο, θα συνεχίσετε να συγκεντρώνετε ε, αρμοδιότητες και να τις ε, δίνετε τελικά σε τεχνοκρατικούς οργανισμούς και όχι στις διοικήσεις και τελειώνω, τελειώνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουρτάσουν. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Πραγματικά αν, καταστρα... αν, αν υπάρξει αναστολή των ταμείων θα ήταν πραγματικά φοβερό. Αλλά είμαστε εδώ για δύο αποφάσεις που συνδέονται με την κυβέρνησή σας. Η πρώτη, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται να μην το θυμάται κανείς, το 2013 έχουμε το μακροοικονομικό αυτό κριτήριο ε, για τα ταμεία. Και εσεί δεχτήκατε αυτό το κριτήριο, δεχτήκατε την επαγγελματική διαδικασία ως κυβέρνηση, το κόμμα σα το δέχτηκε εδώ και σχετίζεται αυτό με τη σημερινή κατάσταση. πέρσι είναι και πολύ κακή δημοσιονομική ε, διαχείριση. Είπατε ότι θα φτάσει 4,6%. Το ίδιο είπατε ε, πριν από μερικά χρόνια και βρεθήκατε εκτό στόχων. Η δημοσιονομική σα διαχείριση και η ε, η φορολογική μεταρρύθμιση τι έκανε τελικά, μείωσε τον προοδευτικό χαρακτήρα ε, της φορολόγησης, μειώθηκαν οι φόροι για του πιο πλούσιου. τελικά για το 2015 είχαμε μείωση ε, των εισπράξεων 1,3 δις. Λίγο πολύ αυτό που σας ζητάνε τώρα δηλαδή. Σεπτέμβριο του 2016, μείωση των εισπράξεων 330 εκατομμύρια. Ε, και μας λέτε τώρα ότι θα πληρώσουν προκαταβολή οι επιχειρήσεις. Ε, μείωση 22,5% έως το Σεπτέμβριο παρουσίαση πράξη για το φόρο επιχειρήσεων. Τι θα κάνετε τελικά, ε, θα σταματήσετε αυτή την ε, μεταρρύθμιση, την, την δημοσιονομική και μπο, είχατε πει ότι θα μειώσετε τους ε, φόρους προεκλογικά. Θα ζητήσετε συγγνώμη γι' αυτό. Ευχαριστούμε και τώρα από την EFTD έχουμε κάποιον όχι, η ΕΝΕΦ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο σύνολο των ερωτημάτων. Πρώτα απ' όλα, ποιο θα είναι το δημόσιο έλλειμμα της ε, ε Ισπανίας για το 2016. Εμείς έχουμε διαπιστώσει ότι η τροποποίηση που κάναμε σε ό,τι αφορά το φόρο επιχειρήσεων σημαίνει ότι και οι εισπράξεις που θα έχουμε για την πρώτη δόση τον Οκτώβριο έχουμε ξεπεράσει τους στόχους μας, την προβολή που είχαμε κάνει εν περιπτώσει. λοιπόν κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η εισπράξη μετά την τροποποίηση του φόρου επιχειρήσεων μπορεί να ξεπεράσει την αρχική μας προβολή που ήταν 830 εκατομμύρια και να είναι γύρω στα 900 εκατομμύρια και το λέω αυτό βέβαια επιφυλακτικά, συντηρητικά. Αν έτσι είναι τα πράγματα και, και αν λάβουμε υπόψη μας και τις ε, δαπάνες, το 4,6% ο στόχος είναι ένας στόχος απολύτως εφικτός. Θεωρούμε ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες να τον πετύχουμε και βεβαίως ανάλογα με το πώς θα κλείσει ο προπολογισμό, ε, αυτός ο στόχος ε, είναι απολύτως εφικτός και μπορούμε και να τον ξεπεράσουμε. Το να βρεθούμε κάτω από το στόχο ε, θα ήταν εξαιρετικά καλό. Θα ήταν εξαιρετικό για τον στόχο του ερχόμενου έτους που είναι 3,1%. Αυτό θα, θα διευκόλυνε την, την προσαρμογή καθώς ε, και θα ήταν καλό να έχουμε και ένα αριθμό ανάπτυξης υψηλότερο από αυτόν ε, που έχουμε εμείς προβλέψει επιφυλακτικά πάντα και συντηρητικά. Η πρόβλεψη της Ισπανικής κυβέρνησης είναι το 2,9% για το 2016 και 2,3% ε, για το επόμενο έτος. Αυτές οι προβολές είναι εξαιρετικά συντηρητικές, έτσι. Όλοι οι αναλυτές, θα δούμε τι θα πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προβολές της αύριο, λένε ότι η Ισπανία ε, θα έχει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3% για φέτος. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε έτσι, θα, έρθουμε με φόρα για το 2017 και ο στόχος του 3,1 ε, μάλλον ο στόχος για το, η προβολή ανάπτυξη 2,3 για το 2017 και αυτή είναι συντηρητική. Μια υψηλότερη ανάπτυξη θα βοηθήσει στο να μειώσουμε και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Έτσι λοιπόν το 4,6 σίγουρα μπορούμε να το πετύχουμε ε, για το έλλειμμα και αυτό σημαίνει ότι το σημείο αφετηρίας για το στόχο του 3,1 του 2017 θα είναι επίσης ε, εξαιρετικό. Τώρα έγινε αναφορά στην, ε, στον τομέα της οικοδομής και της ε, αγοράς εργασίας. Κατά τη διάρκεια ε, της κρίσης χάσαμε περίπου 10 μονάδες από το ΑΕΠ ε, λόγω των οικοδομών. Δηλαδή βυθίστηκε ο κλάδος αυτός και είναι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους η απασχόληση ε, είχε τόσο αρνητική εξέλιξη. Ξέρετε ότι ο τομέα τη οικοδομή ε, είναι εξαιρετικά εντατικό ό,τι αφορά το εργατικό δυναμικό. Όταν πάνε καλά τα πράγματα, δημιουργεί πολλέ θέσει απασχόληση και όταν δεν πάνε καλά, γίνεται το αντίθετο. Και αυτό έγινε στην Ισπανία. 40-50% της ανεργίας στην Ισπανία στην εποχή της κρίσης προέρχεται από την καταστροφή θέσεων εργασία στον τομέα της οικοδομής. Αυτή τη στιγμή ο τομέας αυτός έχει σταθεροποιηθεί και έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ότι μετά από μια προσαρμογή τιμών που ξεπέρασε το 1 τρίτο αυτή τη στιγμή έχουν, έχουν αρχίσει να αυξάνονται και πάλι οι τιμέ μετά από μια μείωση τη τάξη του 33%. Αυτό έχει να κάνει και με την ε, ε, χρηματοοικονομική εξυγίανση βέβαια, διότι συνδέεται η εξέλιξη στις τράπεζε με την εξέλιξη στην τομέα τη οικοδομή, μια και η χρηματοδότηση, τα ανυπόθηκα δάνεια, η χρηματοδότηση των ε, ε μεγάλων εργολάβων σχετίζεται με την τραπεζική δραστηριότητα. Και βεβαίω είχαμε και την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών. Είμαστε μια ανταγωνιστική οικονομία. Είμαστε μια οικονομία όπου οι εξαγωγέ αυξάνονται πάνω από το παγκόσμιο εμπόριο. Είμαστε η οικονομία τη Ευρωζώνη όπου οι εξαγωγέ έχουν το μεγαλύτερο δυναμισμό και αυτό δείχνει την ανταγωνιστικότητα τη ισπανική οικονομία. Τώρα, εργασιακή αγορά, αγορά εργασία, τέθηκε ερώτημα από την κυρία Μπερέ προηγουμένω. Ε, εγώ αυτό που πρέπει να σα πω ότι οι φτωχοί εργαζόμενοι ε, εντάξει, εμείς είχαμε έτσι, υπενθυμίσω, 27% ε, φτωχών εργαζομένων που ήταν άνεργοι. Έτσι. Αυτή είναι η βασική πηγή φτώχειας και ανισότητας. Ιδιαίτερα η ανεργία μακρά διαρκείας. Ε, έχουμε λοιπόν ανακτήσει τα, τις μισές της εργασίας και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Τώρα, η ε, εξέλιξη των ε, μισθών στην Ισπανία αρχίζει σχεδόν σχεδόν να ξεπερνάει ε, τον πληθωρισμό. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό. Σημίζω ότι είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κάποιε θετικέ επιπτώσει ε, σε επίπεδο δραστηριότητα. Ε, αυξάνεται έτσι βεβαίω και η αγοραστική δύναμη. Έγινε μια αναφορά στι δημόσιε διοικήσει. Η προσπάθεια μείωση ε, των δαπανών στο διοικητικό, διοικητικό επίπεδο είναι προφανώς απαραίτητη. Στην Ισπανία έγιναν μεγάλες προσπάθειες. Μπορεί να φαίνονται λίγες, αλλά έγιναν σημαντικές προσπάθειες. Νομίζω ότι αν κάποιος δει τι γίνεται ε, με την δημοσιονομική προσαρμογή στη χώρα μας, διαπιστώνει ότι οι κοινωνικές δαπάνες παραμένουν, διατηρούνται, χάρη στην ανάπτυξη ε, τον, ε, την αύξηση των συντάξεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία, να αποφύγουμε τις ε, επικαλύψεις. Βεβαίως πρέπει να γίνουν πολλά. Όμως, και αυτό είναι προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης, συμφωνήσαμε και με την αντιπολίτευση, να σταματήσει η γύρανση του πληθυσμού, να αντιμετωπίσουμε τη γύρανση του πληθυσμού στα πλαίσια της συμφωνίας του Τολέδο, είναι βασική, βασικό στοιχείο για τη βιωσιμότητα των δημοσίων δαπανών. Τώρα, η προσαρμογή στην Ισπανία. 4,6% ε, λέμε φέτο το έλλειμμα. Ε, και μπορούμε να πέσουμε στο 3,1%. Αυτός ο οικονομικός κύκλος μπορεί να μας δώσει περίπου μία ποσοστία μονάδα. Στη συνέχεια θα πρέπει βεβαίω να πάρουμε για κάποια μέτρα πέρα από την ανάπτυξη που θα μας δώσει 1% για να μειώσουμε το έλλειμμα. Υπάρχει ακόμα μισό μισό του ΑΕΠ, 0,5 του ΑΕΠ. Θα έρθουν σε επαφή με τις, ε, τα πιο σημαντικά κόμματα του Κοινοβουλίου μας. Θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ένα πακέτο μέτρων που θα είναι το κατάλληλο και σε σχέση με τους οικονομικούς μας στόχους και σε σχέση υπό το πρίσμα δηλαδή τη ρευστότητα. Και βέβαια η παραγωγικότητα είναι πολύ σημαντική. Η παραγωγικότητα συνδέεται με την εκπαίδευση, συνδέεται με την έρευνα, την ανάπτυξη και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό το ζήτημα. Το θέμα τώρα της ε, ε φορολογικής ε, μεταρρύθμισης ε, είναι κάτι που εξηγεί την ανάπτυξη της Ισπανίας αυτή η μεταρρύθμιση. Ήταν σημαντική ιδιαίτερα το 2015. Το 2016 βεβαίως δεν είχαμε άλλες μεταρρυθμίσεις αλλά συνεχίζει να έχει την ανάπτυξη πάνω από 3% η ισπανική οικονομία και αυτό σχετίζεται με δύο στοιχεία. Πρώτον, η Ισπανία είναι ανταγωνιστική, όπως άλλωστε δείχνουν οι εξαγωγές της, και δεύτερον, το χρηματοοικονομικό ε, σύστημα της Ισπανίας έχει εξηγενθεί. Ευχαριστούμε. Τελευταίος γύρος από τις ε, ε, επιτροπές Ample Badge Agri. Ο κύριος Φερνάντες πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέτε ότι δεν πρέπει, η δική μας Επιτροπή έχει πει ότι δεν πρέπει να υπάρξει αναστολή των διαδοτικών ε, κονδυλίων για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το Συμβούλιο αποφάσισε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον αποφάσισε να μην τιμωρήσει την Ισπανία. Υπάρχουν, ε, υπάρχει ένα σύνολο κανόνων και ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο και γνωρίζουμε και τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Ισπανία. Με επιχειρήσεις, εργαζόμενους, ε, αλληλείς, νέους, ε, ενώσεις, όσους έχουν προβλήματα φτώχειας. Η αναστολή των διευθυντικών κονδυλίων θα καταστούσε και θα ακύρωνε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια που έχει γίνει από τον Ισπανικό λαό. Επίσης, έπρεπε η Ισπανία να έχει πρόσβαση σε 800 εκατομμύρια ε, ευρώ ως προς την χρηματοδότηση. Δεν μπορεί λοιπόν να ε, προβλέπεται από τη μία πρόσβαση της Ισπανίας και από την άλλη να υπάρχει αναστολή. Μας φαίνεται παράλογο κάτι τέτοιο, μας φαίνεται ε, άτοπο και δεν έχει και κανένα λόγο να πραγματοποιηθεί. Κύριε Υπουργέ, πώς βλέπετε αυτή την πιθανότητα αναστολής. Ευχαριστούμε για την επιτοπή. Έμπλε ο κύριος Γκουτιέρες Πρεγιατού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, μετά την παρέμβασή σας ε, θα ήθελα να σας απαντήσω σε κάποια πράγματα που είπατε για το πώς ε, έγινε αυτή η εξυγίανση, τι είδους θέσεις εργασίας δημιουργούνται, τι μισθούς δίνεται, ε, ποιοι αυξάνονται και ποιοι μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ είμαστε σήμερα διότι η Ισπανία ξεκινάει τη διαδικασία ε, της ενδεχόμενης αναστολής των διαδροτικών πόρων λόγω ε, αύξησης του ελλείμματος. Και αυτό επειδή πέρυσι είχαμε πολύ ε, σημαντικές ε, σημαντικέ αποκλήσει επειδή κάνατε αυτή τη μεταρρύθμιση η οποία ήταν υπέρ των πλούσιων και κατά των φτωχών. Αν δεν είχα κάνει αυτή τη μεταρρύθμιση, δεν θα ήσασταν εδώ σήμερα να δίνετε εξηγήσει. Ε, θα είχατε πετύχει το στόχο ε, του, των Βρυξελών. Δεν είμαι εδώ για να σα κατηγορήσω όμω. Είμαι εδώ για να σα πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σα υποστηρίζει. Η, η σοσιαλιστική ομάδα σα υποστηρίζει. Υποστηρίζει την Ισπανία, όχι εσά. Είμαστε κατά βεβαίω αυτών των ε, όρων που έχουν τεθεί. Το έχουμε πει ε, εδώ και καιρό των μακροπρόθεσμων όρων πρέπει να εφαρμοστεί το άρθρο 23 που λέει ότι αν η Ισπανία προτείνει διορθωτικά μέτρα η διαδικασία κυρώσεων πρέπει να ε, ανασταλεί. Τώρα, ε, το θέμα είναι πώς η Ισπανία θα πετύχει το 0,5% διαθροτικής μείωσης και αυτό πρέπει να γίνει μέσω εσόδων από μια παρέκκληση της δικής σας μεταρρύθμισης μέσω του φόρου των επιχειρήσεων, του φόρου στο κεφάλαιο ή προλογώντα ε, προλογώντας πιο ε, υψηλά εισοδήματα ε, στο φόρο εισοδήματος. θα είναι αυτό δεσμεύστε για κάτι τέτοιο κύριε Ευχαριστούμε για την Επιτροπή Άγκρη, η κυρία Νταγέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η φωνή μου έχει κλείσει κάπως. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω την παρέμβασή μου και να με ακούσετε καλά. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Έχουμε κυβέρνηση στην Ισπανία πλέον. Είστε και πάλι υπεύθυνο ε, των οικονομικών και πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να υποβάλλετε ένα νέο προπολογισμό, ένα νέο προπολογισμό ισορροπημένο που να έρθει να διορθώσει τα λάθη του παρελθόντος τις ανισορροπίες. Δεν μπορεί πάντα οι πιο φτωχοί, αυτοί που φέρουν πιο πολύ, να είναι αυτοί που θα βλέπουν τα δικαιώματά τους να, να συρρυκνώνονται. Οι Ισπανοί ήδη έχουν σφίξει πολύ το ζωνάρι. Έχουν υποφέρει. Είχαν, είχαμε πολύ σημαντικές περικοπές και στα δικαιώματά τους και στην ποιότητα ζωής τους. Ιδιαίτερα τα τέσσερα χρόνια ε, που κυβερνήσατε εσείς δεν τους αξίζουν περισσότερες περικοπές. Καλό θα είναι να εξηγήσετε σήμερα εδώ τα 5,5 δις που σας ζητήσαν να περικόψετε, που, από πού θα τα περικόψετε τον προπολογισμό. Επίσης να σας πω ότι οι αυτόνομες περιφέρειες όπως η Ανταλουσία η δική μου, η Ανταλουσία πέτυχε ε, το στόχο για το έλλειμμα. Δεν μπορείτε λοιπόν να τους κατηγορήσετε. Δεν μπορείτε να τιμωρήσετε αυτούς που έκαναν αυτό το σωστό όπως ε, ε τους Δήμους. Έτσι λοιπόν υποστηρίζω την κυβέρνηση της Ισπανίας η Επιτροπή Γεωργίας είναι κατά της αναστολής των τεχνικών ταμείων αυτό θα ήταν ένα αχρίαστο και άδικο κακό. Ευχαριστούμε για την Επιτροπή ΠΕΣ ο κ. Μάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ για την προσπάθεια που, έχετε, που έχει κάνει όλος ο Ισπανικός λαός να ξεπεραστεί το η κρίση που ήταν ιδιαίτερα έντονη στη χώρα μα. Η Ισπανία είναι ένα πολύ σαφέ παράδειγμα σε ό,τι αφορά τι μεταρρυθμίσει, αλλά και σε επίπεδο ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων απασχόληση και μείωση του ε, ελλείμματος. Για όσου δεν το βλέπουν, τα στοιχεία υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, το να μιλήσουμε για αναστολή των διαδρομικών ταμείων και πάγωμα ε, θα ήταν κάτι που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε, θα ήταν παράλογο. Δεν θα μπορούσαν να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι πολίτε που θα έβλεπαν ότι τελικά η συνταγή της Ευρώπης είναι ε, όταν κάνει κάποιες προσπάθεια το τιμωρούμε. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Ε, δεν υπάρχει κανένας κανόνας άλλωστε που να προβλέπει κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω πολύ μακριά την Ισπανία, από τις Κανάριες νήσους, από μια υπερπεριφερειακή ζώνη, αλλά ιδιαίτερα ευρωπαϊκή, με πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και με μια τεράστια εξάρτηση από αυτά τα ταμεία. Από εκεί λοιπόν και από εδώ εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι δεν θεωρούμε ότι η Ισπανία αξίζει να, να παγώσουν τα ταμεία. Και ένα τέτοιο μέτρο τόσο άδικο δεν πρόκειται να λάβει χώρα. Δεν ήταν κακό για την Ισπανία, θα ήταν ακόμα χειρότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε χρόνο για δύο μόνο κατστιά, ο κύριος Μπαρκασέλ. Ευχαριστώ, Πολλές φορές εμείς έχουμε μιλήσει κατά της αναστολής των διαθροτικών ταμείων προς την Ισπανία για, λόγω του περιβολικού ελλείμματος. Το να κάνει κανείς κάτι τέτοιο θα ήταν καταρχήν άδικο. Άδικο σε σχέση με την προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι Ισπανοί όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης θα ήταν κάτι επιζήμιο όχι μόνο για τα συμφέροντα της Ισπανίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι έρχεται να τροφοδοτήσει τους λαϊκισμούς κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και επίσης διότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ως όργανο κυρώσεων και τιμωρίας σε ό,τι αφορά το υπερβολικό έλλειμμα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να μάθει να κλείνει το ρήμα ε, είμαι ευέλικτο. Χάρη στη μεταρρύθμιση της Ισπανικής κυβέρνησης μπορέσαμε να ανατρέψουμε τους αρνητικούς αριθμούς και στον τομέα της ανεργίας. Βεβαίως πολλά μένουν να γίνουν. Είναι όμως αλήθεια ότι αυτός είναι ο δρόμος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Χώνας Φερνάντες. Δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία που θα ξεκινήσει τώρα, ε, το Σεπτέμβριο ήδη είπαμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να επιβάλλει οποιοδήποτε τέτοιο ε, πάγωμα και τον Αύγουστο το είχαμε πει αυτό είναι αλήθεια ότι η ισπανική οικονομία έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα όμως να μου είχε πει ο υπουργό να γνωρίσει ε, ότι η διάσωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε ε, τη διάσωση του τραπεζικού τομέα, έτσι, ε, και να γίνει αναφορά και στο έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που επιτρέπει ε, να έχουμε ε, πολύ χαμηλά επιτόκια σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή μας. Λοιπόν, είναι Ηράκλειο το έργο μας, εξακολουθούμε να έχουμε πολύ υψηλό, υψηλή ανεργία, έχουμε νέο, νεόπτωχους επίσης ε, πολύ σημαντικούς ε, σε αριθμητικά στοιχεία, δεν πρέπει λοιπόν σε καμία περίπτωση να παγώσουν τα ταμεία. Υποστηρίζουμε λοιπόν την Ισπανική κυβέρνηση, υποστηρίζουμε την Ισπανία, έτσι ώστε να μην υπάρξει οποιαδήποτε κύρωση απέναντι στην Ισπανία. Ευχαριστώ. Please, Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Σημερίζομαι αυτό που είπαν πολλοί σχετικά με την αναστολή ε, των, ε, των ε, ταμείων ως μια απειλή αξιόπιστη. Δεν είναι μια αξιόπιστη απειλή. Το μόνο που θα έκανε κάτι τέτοιο, όχι μόνο δεν θα πετύχαινε την ε, το στόχο, δηλαδή να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα, το μόνο που θα πετύχαινε θα ήταν το αντίθετο. Να μειωθεί ε, να μειωθούν τα φιλοευρωπαϊκά συναισθήματα που υπάρχουν και στην Ισπανία αλλά και στην Πορτογαλία. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε άλλα μέσα, πιο πιστικά, πιο αποτελεσματικά. Πιστεύω πως είναι πολύ καλύτερο να σκεφτούμε ότι μια χώρα όπως η Ισπανία που έχει 100% ε, δημόσιο χρέος, 100% του ΑΕΠ και πρέπει να μειώσει το χρέος αυτό σε ένα σωστό ρυθμό έτσι ώστε να υπάρξουν εγγυήσει ε, σε δημοσιονομικό επίπεδο παρά να έχουμε ε, κανόνες έτσι υπεραπροστευτικούς, απειλητικούς που δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν όπως η αναστολή των διαθροτικών ταμείων ή η επιβολή ενός προστίμου. Έτσι λοιπόν συμμερίζομαι αυτό που είπαν πολλοί από εσά ότι εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Πρέπει να βρούμε άλλα μέσα αποτελεσματικά έτσι ώστε να υπάρχει βεβαίως ε, δημοσιονομική ισορροπία και να το σεβόμαστε αυτό στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης όπου πρέπει να μοιραζόμαστε το ρίσκο και να αποφεύγουμε και τις ανισορροπίες. Τώρα, έγιναν κάποιες ερωτήσεις για τις διαθροτικές περικοπές που πρέπει να κάνει η Ισπανία. Μισό της 100 του ΑΕΠ. Θα πρέπει να το μοιράσουμε αυτό μεταξύ δαπανών, εσόδων. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες επικαλύψεις που μπορούν, να, να εξοικονομήσουμε κάποια χρήματα, αλλά ε, το βασικό είναι να έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης. Να έχουμε ρυθμό ανάπτυξη υψηλό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματο για μια οικονομία σαν την Ισπανική εάν δεν παραμείνει η οικονομική ανάπτυξη. Και αυτό σχετίζεται πολύ περισσότερο με οικονομικέ μεταρρυθμίσει, με την εξυγίανση του χρηματοοικονομικού τομέα, με την αναζήτηση ανταγωνιστικότητα, με τη δημιουργία θέσεων απασχόληση μέσω ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων. Βεβαίω, να γνωρίζω τη σημασία τη ε, τραπεζική εξυγίανση. Βλέπω άλλε χώρε που το 2012 μα έλεγαν α κάναμε αυτό που έκανε η Ισπανία το 12, διότι η Ισπανία τώρα είναι πάνω από ε, στην ανάπτυξη και άλλες δεν φτάνουν στο 1%. Το αναγνωρίζω. Η εξυγίανση των τραπεζών, η διάσωση των τραπεζών ήταν βεβαίως εξαιρετικά σημαντική. Αλλά και οι πολιτικές της ΕΚΤ. Αλλά οι πολιτικές της ΕΚΤ είναι πιο αποτελεσματικές στην Ισπανία από ό,τι σε άλλες χώρες. Οι ροές χρηματοδότησης ε, πάνε, αυξάνονται με διπλάσιους ε, αριθμούς, με, με μάλλον διψήφιους αριθμούς και ένα βασικό στοιχείο, το οποίο είδα προηγουμένω, είδα και μια έκθεση τη ΕΚΤ πρόσφατα, ένα σημαντικό θετικό στοιχείο, πιστεύουμε ότι είναι μια ένδειξη ε, τη θετική εξέλιξη ε, του τραπεζικού τομέα, το κόστο χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το ίδιο με αυτό των γερμανικών τραπεζών για τις γερμανικέ ε, μικρομεσαίε επιχείρησει. Αυτό είναι ένα σαφέ σημείο όπου βλέπουμε πώς ε, στην Ισπανία ο χρηματοοικονομικός τομέας εξηγιάνθηκε και χωρίς ένα εξηγεμένο ε, χρηματοοικονομικό τομέα είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει η οικονομική ανάπτυξη. Ε, Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δοκίνητος. Ήταν πολύ επικοδομητικός ο διάλογός μας και σημαντικό να θυμίσουμε ότι ασχέτως της δικής μας πολιτικής αποτίμησης που μπορεί να διαφέρει ακόμη και αν κάποιοι θέλουν τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα μη σκόπιμη. Ε, παρόλα αυτά, σημαντικό είναι ότι βάσει του κανονισμού, εάν περάσει σε πραγματική δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή μάλλον εάν θεωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ιδέωσες ενέργειες έχουν αναλυφθεί, τότε η νομική υποχρέωση έχει καταπίπτει. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσον θα χρειαστεί να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για τη χρήση αυτού του εργαλείου. το εργαλείο αυτό βέβαια που δεν θα τοποθετηθούμε τώρα για το αν είναι το καταλληλότερο ή όχι. Μας ενδιαφέρει τι δράση έχει αναλάβει η οχι μας ενδιαφερει τι δρασεις εχει αναλαβει η ισπανια προκειμένου να εκπληρώσει τι υποχρεώσει τη βάση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Πρόεδρε, ευχαριστώ, Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ για τι λεπτομερεί απαντήσει που δώσατε, καθώ και για την διαβέβαιωσή σα ότι η Ισπανία βρίσκεται στη σωστή οδό. Ευχαρίστω το ακούμε αυτό. Και τώρα η εικόνα που έχουμε είναι πιο πλήρη για την ανάπτυξη της Ισπανίας και πιο εύκολο, επομένω για μας να λάβουμε μια απόφαση σχετική με τον διαρθρωτικό διάλογο. Ε, επισημαίνω ότι ο ρόλος των επενδυτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε κάθε χώρα μέλος, βεβαίω και στην Ισπανία. Και σας υποστηρίζω απολύτως στις προσπάθειές σας να δημιουργήσετε πλούτο και απασχόληση, την στήριξη του τραπεζικού τομέα, την στήριξη της οικοδομής, την στήριξη όλων των τομέων και βεβαίως και του ρόλου των περιφερειών. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τι εξηγήσει που μα δώσατε και θα έχετε την πλήρη υποστήριξη τη Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτύξεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Dear colleagues, please take seat. Σας παρακαλώ καθίστε αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Καθίστε παρακαλώ. Please, I would like to welcome... Θα ήθελα να απευθύνω το καλό ορίσατε στον Πορτογάλο Υπουργό ε, Οικονομικών. Ε, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ήδη έχουμε εξηγήσει το πλαίσιο του διαρθρωτικού διαλόγου, δηλαδή που προβλέπει το άρθρο 23 του κανονισμού μας και η παρουσία σας εδώ είναι σημαντικό μέρος του διαλόγου αυτού. Επιτρέψτε μου με τα λόγια αυτά να δώσω το μικρόφωνο στη συνάδελφό μου κυρία Μιχαήλοβα, η οποία θα διευθύνει τη συζήτηση στο πρώτο αυτό μέρος. Καλά, μου το επιστρέφει το μικρόφωνο η κυρία Γκουαρτιέ. Επομένως θα διατηρήσω τα ενία τη συζητήσεως και παρακαλώ εσείς κύριε Υπουργέ να ε, λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Μέλη της Επιτροπής Ρέντζε, κυρία Μιχαήλοβα, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής ΕΚΟΝ, κύριε Γκουαλτιέρη, κύριε και κύριοι Ευρωβουλευτές. Ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο για την πρόσκληση του. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναπτύξουμε ε, μία, ε, ένα προβληματισμό για την ενδεχόμενη αναστολή των διευθυντικών ταμείων ε, προς ε, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Έχουμε εκλεγεί έχετε κλεγεί μάλλον άμεσα από τους πολίτες, οπότε έχετε την απαραίτητη νόμιμοποίηση για να κρίνετε ως σώμα τέτοιου είδους καταστάσεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικός ο διαθωμένος διάλογος μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Επιτροπής αυτή η διαδικασία δείχνει τον κεντρικό χαρακτήρα και τις αυξανόμενες αρμοδιότητες του Ευρωκοινοβουλίου στα πλαίσια του ευρωπαϊκού θεσμικού διακανονισμού και πλαισίου. Χαιρετίζω λοιπόν αυτό το ρόλο. Για να αρχίσουμε τη συνεισφορά μας αυτό το διάλογο θα ήθελα να τονίσω την ε, σημασία των έω τώρα εκπεφρασμένων θέσεων από το Ευρωκοινοβούλιο επί του θέματος ε, όλες ιδιαίτερως στο πλαίσιο των πρόσφατων ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν και οποία αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να σεβαστούμε την πολιτική συνοχή, εντό τη οποία τα διευθυντικά ταμεία έχουν καθοριστικό ρόλο, όπω και την ε, χρηστή οικονομική διακυβέρνηση. Αυτόν τον, ε, μάλλον τον Σεπτέμβριο, έστειλα επιστολή προ τα μέλη της, ε, των διαφορών επιτροπών σα, εξηγώντα γιατί η Πορτογαλική κυβέρνηση δεν συμφωνεί και δεν θεωρεί ότι υπάρχει λογική στην ενδεχόμενη αναστολή των διευθυντικών κομπιλιών και των επενδυτικών επενδυτικών ταμείων, των κονδυλίων των επενδυτικών ταμείων προ την ε, Πορτογαλία. Τα επιχειρήματα που αναπτύσσονται σε αυτή την επιστολή θα πρέπει να συνδυαστούν με την επιστολή που απεστάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των κυρώσεων. Όπω γνωρίζετε, τον Αύγουστο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΚΟΦΗΝ αποφάσισαν ομοφόνω να κυρώσουν ε, με πρόστιμο την ε, έλλειψη ε, πραγματικής δράσης στην περίοδο 2013-2015, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του λαού της Πορτογαλίας και τη συμφωνία ε, που ε, θα πετύχει πετύχαινε η πορτογαλική κυβέρνηση για την τωρινή κατάσταση και τη μελλοντική. Η συζήτηση συνεχίζεται και η συλλογιστική βεβαίω οδήγησε το. Ε, η συλλογιστική οδήγησαν το Επιτροπή και το Συμβούλιο να ακυρώσουν την επιβολή ποινή. Βεβαίω, ε, συζητούμε μία ενδεχόμενη ποινή που θα ήταν ουσιαστικά ποινή κατά των πολιτών και των επιχειρήσεων τη Πορτογαλία και όχι τη κυβέρνηση. Κάτι που θα κατέστρεφε την εμπιστοσύνη των Πορτογάλων στην Ευρώπη σε μία ένωση όπου μετράνε οι πολίτε. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί και γι' αυτό δεν θα συμβεί. Επιτρέψτε μου να αναπτύξω με σύντομα επιχειρήματα, γιατί αυτή η αποφάση δεν θα είχε καμία οικονομική ή πολιτική ε, λογική. Σε αυτή τη διαδικασία η πολιτικη λογικη σε αυτη τη διαδικασια η επιτροπη στο πλαίσιο του κανονισμού 1303-2013, θα πρέπει να λάβει υπόψη όλε τι ε, σκόπιμε πληροφορίε, όπω και τον αντίκτυπο αυτή τη ενδεχόμενη αναστολή στην ε, κοινωνία και την οικονομία με ε, την αρχή τη αναλογικότητα να εφαρμόζεται στον αντίκτυπο των ενδεχόμενων αποφάσεων. Εδώ ε, υπάρχει το επιχείρημα που λέει ότι απλώ συζητάμε το ενδεχόμενο αναστολή ε, των συμφωνιών. Κάτι όμω που μπορεί να έχει άμεσο ε, αντίκτυπο στι εκταμιεύσει. Μια καθυστέρηση από το πραγματικό αντίκτυπο μια τέτοια αναστολή ήδη θα έστελνε μια σειρά από αρνητικά μηνύματα. Και θα ήταν πολιτικό τιμωρητικό αυτό τη στιγμή που η Πορτογαλία ετοιμάζεται να ξεκινήσει η διαδικασία επί ε, υπερβολικών ελλημάτων. Οι πορτογαλικές και οι ευρωπαϊκές αρχές ήδη έχουν κάνει πολύ επικοδομητικό διάλογο τον τελευταίο χρόνο και δεν θέλουμε να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών εντό είτε εκτό τη χώρα, ούτε να καθυστερήσει να ακυρωθεί η εκπόνηση, η εκτέλεση έργων και να χαθούν νέε θέσει εργασία ε, δυσκολεύοντα την οικονομική ανάπτυξη. Το Συμβούλιο αποφάσισε να μην επιβάλλει πρόστιμο στην Πορτογαλία βάσει μετά την πρωτοδισεκτική εξέταση των ε, κριτηρίων που έχουν οριστεί στον κανονισμό 1173 του 2011. Το Συμβούλιο αναγνώρισε ότι παρόλο που επιτεύχθησαν ορισμένοι από του στόχου του προπολογισμού, η χώρα έχει καταβάλει τεράστια προσπάθεια. Η Πορτογαλία μείωσε το δημόσιο έλλειμμα από 8,6% του ΑΕΠ το 2010 σε περίπου 3% το 2015, ε, χωρί να λαμβάνονται υπόψη καν τα προσωρινά μέτρα. Όπω συμφωνήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόστηκαν διαδοτικέ ε, μεταρρυθμίσει, των οποίων αντίκτυπο έχει αρχίσει να παίρνει ήδη να, μόλις τώρα να παίρνει σάρκα και ωστά. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές απαιτούν ε, οικονομική ανάπτυξη για να υλοποιηθούν πλήρως και η έγκρισή τους σε μια περίοδο ύφεση Ένωσης ότι υπήρξε τεράστιο ε, κοινωνικό κόστος το οποίο έλαβαν όλοι οι Πορτογάλοι πολίτες. Αυτό το κόστος σημαίνει υψηλή ανεργία, περίπου 17%, μεγάλης διάρκειας, αλλά και μεγαλύτερο κύμα ε, μετανάστευσης εκτός της χώρας από τότε που άρχισε να έχει χώρα δημοκρατικό πολίτευμα εδώ και 40 χρόνια. Οι διαστάσεις αυτής της προσπάθειας και των συνεπειών της αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια και μετά το πρόγραμμα προσαρμογής. Να προσθέσω ότι πέραν της ακύρωσης του επιβολής προστήμου το Συμβούλιο ε, εφάρμοσε μέτρα, ε, έθεσε μάλλον στόχους για τον προπολογισμό το 2016. Έλλειμμα 2,5% του PIB και διατήρηση του ΑΕΠ και διατήρηση της προσπάθειας για την ε, διευθυντική προσαρμογή. Η πορτογαλική κυβέρνηση υποσχέθηκε να πετύχει αυτούς τους στόχους και οι εταίροι μας στο Eurogroup επένεσαν αυτές τις προσπάθειες. Η εκτέλεση του προπολογισμού θα επιτρέψει να φτάσουμε τους στόχους που συμφωνήθηκαν με τους Ευρωπαίους εταίρους. Το 2016 η πορτογαλική κυβέρνηση πρόκειται να υποβάλει ένα μεγαλύτερο πρωτογενέ πλεόνασμα 1,9% και το μικρότερο δυνατό ονομαστικό έλλειμμα 2,4% των τελευταίων 40 χρόνων. Η διαρθρωτική μα προσαρμογή θα αυξηθεί κατά 0,2 ποσοστιαίε μονάδε. Η Πορτογαλία επιτέλου θα βγει από την διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο πέραν των τεράστιων οικονομικών και κοινωνικών θυσιών, σε μια εποχή που έχουμε να εκπληρώσουμε στόχους στον προπολογισμό, τέτοιου είδου κυρώσει δεν θα γίνονταν ε, κατανοητέ ούτε από του πολίτε τη Πορτογαλία, ούτε από του υπόλοιπου πολίτε τη Ευρώπη. Για του οποίου η Ευρώπη είναι ακόμη ένα χώρο συνεργασία, κοινωνική αλληλεγγύη και οικονομική ευημερία. Α ε, δούμε όμως πώς έχει στην πραγματικότητα η κατάσταση η διαδικασία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αντικατοπτρίζει μια υποτιθέμενη έλλειψη πραγματική δράση στην περίοδο 2013-2015. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, η Πορτογαλία εφάρμοσε μεταρρυθμίσει και οι Πορτογάλοι ε, κατέβαλαν τεράστιε τιτάνιε προσπάθειε. Το γνωρίζουμε αυτό. Σήμερα, επίση, γνωρίζουμε ότι η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματο ε, πρόκειται να οδηγηθεί σε αίσιο πέρα. Και αυτό θα γίνει με τρόπο βιώσιμο. Ο προπολογισμό του κράτου για το 2017 ε, δίνει συνέχεια στην στρατηγική τη ε, ε, Σταθεροποίηση του προπολογισμού στα πλαίσια του ελέγχου των δαπανών, τη δημοσιονομική ε, σταθερότητα και τη προώθηση τη ε, ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή. Η προώθηση λοιπόν τη συμμετοχική ανάπτυξη είναι καθοριστική σημασία. Η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 2%, η ανεργία έχει πέσει στο 15% περίπου, δίνοντα ένα ποσοστό ανεργία 10,8%. Μάλλον έχει πέσει κατά 15% σε σχέση με πέρσι. <clears throat> αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να, να καλέσουμε τι πολιτικέ μα συμφωνίε, από η απάντηση είναι όχι. Από την οικονομική λοιπόν σκοπιά, αυτού του είδου η αναστολή θα ήταν αντιπαραγωγική. Τα ε, κονδύλια της, ε, των Δυτικών Ταμείων είναι καθοριστική σημασία. Στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματο Μεταρρυθμίσεων, η απάντηση στι αναχώρασει τάση και ο τρόπο που εκτελέστηκαν επενέθηκε από την Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε περισσότερη ανταγωνιστικότητα και σύγκληση τη πορτογαλική οικονομία με την ευρωπαϊκή τα ευρωπαϊκά ταμεία μπορούν να στηρίξουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Είναι το 78% των δημόσιων επενδύσεων. Μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2016 η Πορτογαλία έλαβε ένα ε, εκατομμύριο ευρώ, το οποίο προσωπεί 5% του συνολικού ε, κονδυλίου για την Πορτογαλία μέχρι το 2020 και περίπου το διπλάσιο του ευρωπαϊκού μεσοόρου που είναι 3%. Αυτό δείχνει τη σημασία των κονδυλίων της για τι πορτογαλικέ και ευρωπαϊκέ επιχειρήσει που λειτουργούν στην Πορτογαλία. Η αναστολή λοιπόν αυτή έχει τεράστιο αντίκτυπο στην οικονομική μα ανάκαμψη. Η οικονομική κατάσταση τη Ευρώπη δημιουργεί πολλέ αβεβαιότητε μετά τα αποτελέσματα του Βρετανικού δημοψηφίσματο. Πορτογαλικέ επιχειρήσει θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αγορέ που έχουν άλλε δυσκολίε στην Αφρική και στην Λατινική Αμερική. Με μεγάλες επιβαρύνσει σε μια περίοδο οικονομικής ανάπτυξης. Να προσθέσω ότι η αναστολή των πολιτικών συμφωνιών για τα διευθυντικά ταμεία θα έθετε να αμφιβόλο την ανάκτηση της εμπιστοσύνη μας και θα αυξήσει τα προβλήματα που έχουμε από την έλλειψη ε, ανάπτυξης, πλούτου και ε, την, ε, την οικονομική πρόοδο της χώρας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσον δεν υπήρξε πραγματική δράση για την περίοδο 2013-2015 και να μην ακυρωθούν οι προ... παρελθούσες προσπάθειες ε, της Πορτογαλίας για, την, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση διευθυντικών μεταρρυθμίσεων με τόσο μεγάλο κοινωνικό κόστος, ενώ καταφέραμε το μεταξύ να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να ανακτήσουμε ένα μερίδιο της απασχόλησης και να προωθηθεί η επένδυση για την Πορτογαλία. Για να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να εκφράσω την άποψή μου τον καθοριστικό ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου σε σχέση με τα όσα έχει ε, με πει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναστολή των διευθυντικών κονδυλίων θα είναι τελείω ε, ε, ασύμβατη με την απόφαση να μην επιβληθεί πρόστιμο και θα δημιουργήσει τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Πέραν αυτού, θα απομακρύνει κι άλλο του πολίτε από το ευρωπαϊκό εγχείρημα, το Ευρωκοινοβούλιο, θα πρέπει να ε, χρησιμοποιήσει τη δημοκρατική του δυνατότητα να ασκήσει επιρροή, ώστε να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην επιβάλλει ε, αυτού του είδου, ε, να μην λάβει αυτού του είδου την απόφαση και να μην αναστείλει τα κονδύλια. Αυτό ε, δεν, θα πρέπει να είμαστε δέσμοι του πνεύματο και του γράμματο του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει μια συνετή εφαρμογή των υπαρχόντων κανόνων. Διότι όλοι, ε, το σύνολο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων συμπεριλαμβανομένων, θα πρέπει να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, όχι να το θέτουμε ένα αμφιβόλο. Η Πορτογαλία συμμετέχει στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και με βέβαια το Ευρωκοινοβούλιο θα καταφέρει να αναγνωρίσει την δέσμευση του πορτογαλικού λαού να είναι ε, ένα ενεργό μέλος αυτής της προσπάθειας της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχίζουμε πρώτα με την Επιτροπή Οικονομικών. Πρώτο ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα ενώπιόν μας για να απαντήσετε στα πλαίσια του διαθετικού διαλόγου και έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Στο κατατεθειμένο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 θεωρείτε ότι θα έχετε οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 1,5% για τη χώρα σας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ωστόσο, η, αναμονή, αναμενόμενη ανάπτυξη είναι πολύ χαμηλότερη. Για την Ισπανία προβλέπουν 2,5% και νομίζω ότι είναι σημαντική διαφορά και παρόλο που και οι δύο οικονομίες παραδοσιακά είναι στενά συνδεδεμένες. Με ενδιαφέρει πώς εξηγείται τις διαφορές αυτές και αν ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πορτογαλικές εξαγωγές εξαρτώνται από λίγους τομείς και κατευθύνονται και σε λίγες μόνο χώρες, Αγγόλα, Βραζιλία και εν μέρη Κίνα. Για να λάβετε τα αναγκαία, μέτρα θα πρέπει η Πορτογαλία να συνεχίσει τις προσπάθειες για εξυγίανση του εθνικού προϋπολογισμού της. Γιατί τώρα Ωστόσο, μέσα σε μια τέτοια κατάσταση κατεβάζεται και πάλι στο δημόσιο τομέα τις ώρες εργασίας από 40 εβδομαδίως σε 35. Κάτι που μειώνει την ανταγωνιστικότητα και αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες. Ευχαριστώ κύριε Μπερές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κατανοείτε την σημασία του διαρθωτικού διαλόγου και τον σημαντικό θεσμικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως πλαίσιο συζητήσεων. Η αξιοπιστία του διαρθρωτικού διαλόγου βασίζεται επίσης και στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι και φίλοι μας Ισπανοί και Πορτογάλοι που παρεμβαίνουν στην συζήτηση αυτή. Εξού και η σημασία των παρεμβάσεων των συντονιστών και υπό την ιδιότητά μου ως συντονίστριας θα ήθελα πρώτα να σας συγχαρώ για, την, για τις προσπάθειες που έχετε κάνει για την κατάθεση του σχεδίου προϋπολογισμού 2017 αλλά όταν ε, ερωτήσαμε τους επιτρόπους είχαμε αναφερθεί ήδη στον κίνδυνο η περίοδος αβεβαιότητος που αρχίζει έστω και με την υπόθεση αναστολής των πληρωμών των διαθετικών ταμείων να βαρύνει την πορτογαλική οικονομία. Δηλαδή, λόγω της σημασίας των επενδύσεων που προέρχονται από την κινητοποίηση των διαθετικών ταμείων, θεωρείτε ότι ήδη υπάρχει επίπτωση στις επενδυτικές αποφάσεις στη χώρα σας. Επίσης, επιμείνατε στην ομιλία σας στην ανάγκη να δοθεί τελική μορφή στην ε, πολιτική ανάκαμψη και πέραν από την ε, μία αναστολή των διαρθρωτικών ταμείων. Υπάρχουν κάποια μέτρα, ένα, δύο, τρία μέτρα, τα οποία σας φαίνονται απολύτως απαραίτητα. Για παράδειγμα, για το επόμενο ε, ε, σχέδιο επενδύσεων, το λεγόμενο σχέδιο Juncker. Σας ευχαριστώ. για, για τους φιλελευθέρους, Σομπον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Υπουργό για την παρουσία, παρουσία του. Μιλάμε για πολλά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Εσείς ε, δείξατε το πόσο παράλογο, γκροτέσκο θα ήταν να επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο. Στην Πορτογαλία ακόμα περισσότερο, διότι από τα στοιχεία που ε, είδα, ε, εσείς εξετάσετε πολύ περισσότερο για τις επενδύσεις σας στις δημόσιες ε, από τα ε, τα μία τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή θα ήταν οι επιπτώσεις ε, πραγματικά υπερβολικά αρνητικές για σας. Τι θέλω να πω. Έχετε βεβαίως στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ότι δεν πρέπει να συμβεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχει νόημα ε, και θα τιμωρήσουμε έτσι μια χώρα που είναι κάπως αδύναμη που κάνει προσπάθειες, θα την μια κακή εικόνα. Το πρόβλημα βεβαίω υπάρχει και στην περίπτωση της Πορτογαλίας είναι πρόβλημα αυτό το έλλειμμα διότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ε, ε το χατηρισμό του χρέους και αυτό δημιουργεί προβλήματα μετά. Και, και κάτι άλλο, να πούμε ότι κάναμε λάθος παίρνοντας τέτοια μέτρα τιμωρητικά. Είναι ε, πραγματικά παράλογο να παίρνουμε μέτρα τα οποία έχουν σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις. Το να προβλεφθούν δηλαδή τέτοια μέτρα όπως ε, η αναστολή ε, ταμείων πρέπει να βρεθεί κάποιο άλλο σύστημα. Ευχαριστούμε ο κύριος Βιέγκας για την ΚΟΕ. Είναι εδώ. Παρακαλώ, εδώ είστε. Έχουμε μία θέση επί της αρχής κατά της οικονομικής διακυβέρνησης, κατά της μικροοικονομικής ερεσιμότητας και όλα αυτά τα εργαλεία υποδούλωσης της εθνικής κυριαρχίας των κυβερνήσεων. Δια, γι' αυτό είμαστε τελείως κατά της δυνατότητας της ενδεχόμενης αναστολής ε, των διευθυντικών κονδυλίων προς την Πορτογαλία. Το νομικό πλαίσιο θα αποτελέσει φραγμό στην ανάπτυξη και την ίδια την συνοχή που υποτίθεται ότι είναι η θετική στόχη αυτής της διαδικασίας. Πρέπει το πρόβλημα αυτό να τεθεί επιτάπητος. Ιδίως στο επίπεδο του Συμβουλίου, ιδάλλως, μπορεί να αντιτρέξουμε τον κίνδυνο να παραταθεί ένας απαράδεκτος εκβιασμός. Μια κρίση η οποία θα προκύψει αναγκαστικά στο άμεσο μέλλον. Ταυτόχρονα αντιπαραβάλλουμε την ανάγκη να προβλεφθούν επιπλέον μέτρα για να ξεπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, ιδίω σε επίπεδο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώ αυτό ο προπολογισμό βρίσκεται σε φθήνουσα απορία ε, με τιμωρητικές συνεχώς περικοπές. Γι' αυτό, ε, ενώ προτείνεται βοήθεια στις χώρες που έχουν πληγεί από το πρόγραμμα της Τρόικας, που έχει επιβάλει την πολιτική της λιτότητας και έχει δημιουργήσει τον φαυλοκύκλο της φτώχεια και της οικονομικής υποβάθμισης, ε, με τι εθνεί επενδύσει στα κράτη-μέλη μέσω του προγράμματο Juncker για την καλύτερη υποτίθεται κατανομή των επενδύσεων για να ξαναρχίσει η ανάπτυξή μα, αυτέ είναι πτυχέ γενικότερε που δεν μπορούμε να με τι βλέπουμε όταν σκεφτόμαστε το σημερινό σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στα επίπεδα τη ευρωπαϊκή ε, ολοκλήρωση. Ευχαριστούμε κύριο Σουρτασούν. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον ε, Πορτογάλο Υπουργό για την παρουσία του εδώ σήμερα, να του πω ότι εμεί παρακολουθούμε στενά την πολιτική που ακολουθεί. Εμείς ε, βεβαίω είμαστε κατά του παγώματος των ταμείων. Θα ήταν εξαιρετικά άδικο σε μια στιγμή κατά την οποία η Πορτογαλική κυβέρνηση παίρνει μέτρα τα οποία είναι σημαντικά. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα μέτρα που παίρνετε σε φορολογικό επίπεδο. Η πρόταση για το φόρο ε, και κληρονομιά δημιουργεί μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη. Ο νέος φόρος ε, για ε, τα ποτά με πολλά ζάχαρα. Ε, πραγματικά όλα αυτά τα μέτρα που παίρνετε για να μπορέσει να αντιστραφεί αυτό που υπέφεραν οι Πορτογάλοι τόσα χρόνια. Να σας πω λοιπόν ότι εμείς φυσικά και θα σας υποστηρίξουμε όταν θα υποβάλλετε τα μέτρα αυτά και θεωρούμε ότι σαφώς δεν μπορούμε παρά να αρνηθούμε τέτοιου είδους μέτρα εις βάρος σας. Ευχαριστούμε, Διευθυντή, δεν για τους μη γεραμένους κ. Μάλετιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό Χθες ο επικεφαλής του Eurogroup είπε σαφέστατα ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση του πορτογαλικού χρέους. Έτοιμα που είχατε καταθέσει την προηγούμενη εβδομάδα και εκ μέρους του Eurogroup απέρριψε οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάρθρωση του πορτογαλικού χρέους διότι είπε ότι η Πορτογαλία μπορεί να εξυπηρετήσει το ίδιο της το χρέος. Δεν ακούμε την ίδια βεβαιότητα για την Ελλάδα και ούτε θέλουμε να συγχύουμε εδώ στην Πορτογαλία με την Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται σε πρόγραμμα ε, οικονομικής προσαρμογής, ενώ η Πορτογαλία κατάφερε υπό την προηγούμενη κυβέρνηση να εξέλθει από το παρόμοιο πρόγραμμα, άρα δεν βρίσκονται στην ίδια θέση οι δύο χώρες. Επίσης και η Πορτογαλία έχει μεγάλο δημόσιο χρέος, αλλά και η Ιαπωνία και άλλες χώρες έχουν μεγάλο δημόσιο χρέος. Η αίτησή σας για αναδιάθρωση του χρέους θέτει και το ερώτημα αν όντω η Πορτογαλία ακολουθεί σωστά τις πολιτικές τη. Πώς λοιπόν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι και βέβαιοι ότι οι πολιτικές σας έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και ότι οι αναλύσει σας βασίζονται στις σωστές υποθέσεις. Και εάν το Eurogroup συμφωνεί με την Πορτογαλική κυβέρνηση για το χρέο και για την βιωσιμότητά του. Ευχαριστώ. Τα Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ Οικονομικών, σήμερα για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται ότι η θέση πλειοψηφία αυτού του Κοινοβουλίου είναι σαφώ κατά τη αναστολή των κονδυλίων. Διότι η αναστολή αυτή θα είναι και άδικη και δυσανάλογη και αντιπαραγωγική. Όμω, βάσει των όσων μα είπατε σήμερα, μάθαμε ότι πέραν όλων αυτών η αναστολή των κονδυλίων θα ήταν και παράλογη. Η Πορτογαλία δεν χρειάζεται κίνητρα για να συμμορφωθεί με του κανόνε. Για τον απλό λόγο ότι η Πορτογαλία ήδη ακολουθεί πιστά τους κανόνες του ελλείμματος του προπολογισμού 4% φέτος, λιγότερο ακόμη του χρόνου, με προπολογισμό που έχει υποβάλει η κυβέρνησή σα, που θα επιτρέψει ω του χρόνου να έχουμε μεγαλύτερο πρωτογενέ πλεόνασμα στον προπολογισμό και μάλιστα το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρωζώνη. Είναι τόσο παράλογο λοιπόν αυτό, που τίθεται το εξή ερώτημα, Υπουργέ. Γιατί γίνεται μια τόσο παράλογη συζήτηση και κρατάει και τόσο καιρό. Δεν είναι σημαντικό επιτέλους να μπει μια τελεία και μια παύλα σε όλο αυτό το θέμα. Να θυμίσω ότι η απόφαση του Συμβουλίου για την υποτιθέμενη μη ανάληψη πραγματικών μέτρων την ε, εκτέλεση πραγματικής δράσης μέχρι, το χρόνο, το, μέχρι τον φετινό Ιούλιο θα πρέπει να ληφθεί ε, κάποια στιγμή τον Νοέμβριο. Κρατάει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, Υπουργέ. Πλήττεται εντωμεταξύ η πορτογαλική οικονομία, δημιουργεί ένα κλίμα βεβαιότητα και ανασφάλεια. Και επιτέλου, μια και καλή, θα πρέπει να μπει μια τελεία σε όλη αυτή τη συζήτηση για την αναστολή των διευθυντικών κονδυλίων, η οποία είναι παράλογη, άδικη και τελείω αντιπραγωγική. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε και κύριοι Η πορτογαλική οικονομία αναπτύσσεται με τρόπο βιώσιμο τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια του 2016 η ανάπτυξη αυτή έχει επιταχυνθεί. Τα τριμηνιαία ποσοστά είναι υψηλότερα και μάλιστα κάθε φορά και περισσότερο και αυτή η ανωδική πορεία της ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας. Για την αναθέρμανση, την ανάκαμψη της οικονομίας και για να διατηρηθεί αυτό που παρατηρούμε στην αγορά εργασία. Στην ομιλία μου ανέφερα ότι τα προσφατότερα δεδομένα ανάπτυξη για την ε, ε, απασχόληση στην Πορτογαλία δίνουν 2%. Όταν μιλάμε για την κοινωνική ασφάλιση, ε, φτάνουμε σε ακόμη μεγαλύτερα επίπεδα. Έχουμε ανάπτυξη 3% σε σχέση με τον αριθμό των μισθωτών και των όσων είναι είναι εγγεγραμμένη στην ε, κοινωνική πρόνοια της Πορτογαλίας σε σχέση με πέρσι. Αυτό δείχνει ότι οι επισφαλείς θέσει πέφτουν τους τελευταίους μήνες, ε, θα πέσουν κι άλλο κατά 10%. Αυτό λοιπόν ενισχύει την δυναμική άνοδο της πορτογαλικής οικονομίας. Η μεγαλύτερη διαφορά στην οικονομική ανάπτυξη που έθεσε και σε σχέση με την Ισπανία που έθεσε και ο κύριος Μπάλτς έχει να κάνει με το χρηματοοικονομικό σύστημα ως παράγοντα ανάπτυξης. Η ισπανική οικονομία βασίζεται περισσότερο με κεντρικότερο τρόπο στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η πορτογαλική οικονομία πολύ λιγότερο. Και μάλιστα αυτή η κυβέρνηση έλαβε τις αποφάσεις στο τέλος της περασμένης όταν έλαβε, ανέλαβε μάλλον το καθήκοντα τη στο τέλο τη περασμένη χρονιά, αποφάσισε ουσιαστικά να σταθεροποιήσει το χρηματοοικονομικό σύστημα με πολλά μέτρα προ αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να μπορέσουμε και αυτός ο παράγοντας ανάπτυξης να μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και να ανακάμψουμε ακόμη δραστικότερα. Οι εξαγωγέ φέτο στην Πορτογαλία έχουν υποστεί τον σοβαρό αντίκτυπο των όσων έχουν συμβεί, όμως υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή μάλλον υπάρχει ένα ευρύτερο πρόβλημα που αφορά όλες μας τις οικονομίε σε σχέση με τις εξωτερικές αγορά. Ήταν μειωμένο βέβαια, ήταν μειωμένο το βάρος ε, αυτό στις δικές μας εξαγωγές, λόγω, με τη, λόγω χάρη με τη Βραζιλία κατά 1% ή την Αγγόλα 3-4%. Αυτή ήταν η βαρύτητά του στο σύνολο των εξαγωγών μα. Πέρσι όμω είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στην δυναμική πορεία τη ανάπτυξη. Όμω δυστυχώ για διαφορετικού λόγου η ανάπτυξη αυτή αυτή τη στιγμή δεν είναι επαρκή. Οι πορτογαλικέ επιχειρήσει παρόλα αυτά έκαναν κάτι πολύ σκόπιμο. Κατήφθηναν την παραγωγή του σε νέε αγορέ κέρδισαν ε, μερίδια της αγοράς λόγω χάρη σε αγορές πολύ οριμότερες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η, ανά, η εξέλιξη των εξαγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2016 έχει ξεπεράσει την αύξηση των εισαγωγών προς αυτές τις χώρες. Δηλαδή οι πορτογαλικές επιχειρήσεις καταφέρνουν να περάσουν σε μια διεθνή διάσταση και να κερδίσουν αγορές που δεν είχαν πριν. Έτσι ανταποκρίνονται στα οικονομικά πλήγματα. Αναμένουμε λοιπόν ακριβώς η οικονομία μας να επωφεληθεί. Αυτό συνέβη στην πορτογαλική οικονομία ως προς την εξυγίανση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την πορτογαλική οικονομία και η κυβέρνησή μας έχει πάρει πολύ σοβαρά αυτό το ρόλο και όλα αυτά τα ζητήματα. Ως προς την εξυγίανση λοιπόν του προπολογισμού είναι προτεραιότητα. Οι συμβιβασμοί, οι συμφωνίε που πετέχθηκαν σε το Eurogroup είναι ε, κάτι που έχουμε εκπληρώσει ω προ την εξηγένεια του υπολογισμού. Θα φυγούμε από τη διαδικασία του προβολικού ελλείμματο, που είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα ορόσημο για την πορτογαλική οικονομία φέτο. Και το σύνολο μέτρων που έχουμε εγκρίνει στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας τίνουν να μας οδηγήσουν ακριβώς στο να ξεφύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Ο δημόσιος τομέας στην Πορτογαλία πέρασε μια περίοδο πολύ μακρά και δύσκολη, περίοδο προσαρμογής. Οι μισθοί ε, έχουν μείνει ίδιοι από το 2009. Από το 2006 δεν υπάρχουν ε, ιδιαίτερες εξελίξεις στη δημόσια και η αλλαγές που έχουμε επιφέρει στο υπόλοιπο σύστημα της χώρας επηρεάζουν και τη μηχανή της δημόσιας διοίκησης. Έτσι ευνοούνται και αλλαγέ όπω αυτέ που ανέφερε ο κύριο Ευρωβουλευτή, διατηρώντα όμω του περιορισμού στον προπολογισμό, ε, τι περικοπέ αυτέ που είναι τελείω σαφεί, προκειμένου να υλοποιηθούν σωστά τα μέτρα. Είναι βέβαια αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για την ε, πορτογαλική οικονομία, όπω είπε και η κυρία Μπερέ, όμω ο και ο κύριο Θάλμπα μα είπε ότι είναι σημαντική η αξία των κονδυλίων. Να μην ξεχνάμε λοιπόν την ιδιαίτερη σημασία των κονδυλίων για τι δημόσιε επενδύσει και τι ιδιωτικέ στην Πορτογαλία. Μια οικονομία που έχει, βρίσκεται σε έναν ε, θετικό κύκλο ανάπτυξης, ξέφυγε από, τις αρνητικές, ε, από τα αρνητικά στάδια πολύ πρόσφατα και αυτά πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για την οικονομία μας. Η ευρωπαϊκή αφοσίωση της χώρας μας ομοφόνος συζητιέται και είναι αποδεκτή στο εθνικό επίπεδο. Έχουμε φτάσει να απορρίψουμε προκαταρκτικά τουλάχιστον οποιαδήποτε κουβέντα Μάλλον έχουμε ε, απορρίψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εξηγένσης του, της αναδιάρθρωσης του χρέους για το 2017 έχουμε προβλέψει τα απαραίτητα μέτρα για την ε, ε, εξυγίανση του χρέους ώστε να πάψει να βαρύνει την οικονομία μας. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας και είναι μια τιτάνια προσπάθεια ε, στην οποία παραμένει αφοσιωμένη η χώρα μας. Η δυναμική λοιπόν ανάπτυξη που ελπίζουμε να έχουμε και με την ενίσχυση των κοινωνικών κονδυλίων και με την προσπάθεια που θα ε, κάνει η κυβέρνηση στη διάσταση των επενδύσεων, όλα αυτά μπορεί να επηρεαστούν και να περιοριστούν εξαιρετικά εάν προχωρήσουμε σε αυτή την αναστολή. Εάν δηλαδή γίνει πραγματικότητα. Το να συμμορφωνόμαστε με τους κανόνες όπως είπε και ο, ο βουλευτής κύριος ε, Περέιρα είναι θέμα ε, επιλογής πολιτικής της κυβέρνησης της Πορτογαλίας. Είναι προφανές όταν, ότι όταν ε, μήνα το μήνα, έκθεση την έκθεση, όπως είπατε, αυτά τα ερωτήματα να, να ανακύπτουν, προφανώς σέρνονται οι δυσκολίες που έχουμε κι εμείς να υλοποιήσουμε αυτή τη στρατηγική. Και προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο. Κλείνω εδώ με την απάντησή μου ότι η Πορτογαλία είναι δεσμευμένη στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και προφανώς του στόχους που αρμόζουν σε αυτό το πλαίσιο. Πρόεδρος Γκουαλτιέρη, ευχαριστώ πολύ εσείς τώρα κυρία Μιχαήλωβα. Θα συνεχίσουμε τώρα με, την, με τον δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Πρώτος εσείς κύριε Βανίστελ Ρόι, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα, επιθυμώ να πω ότι ο παρόν διάλογος που περιλαμβάνει στον κανονισμό αποδίδει αποτελέσματα. Είναι καλύτερα να συνομιλούμε και να ακούμε οι μεν δε παρά να μιλούμε ημέν για τους δε και να λαμβάνουμε μόνο μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ λοιπόν δημιουργείται μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Το δεύτερο είναι αυτό που βλέπω, ότι δηλαδή και εσείς είστε πολύ θετικό σχετικά με την πολιτική συνοχή και σας ευχαριστώ πολύ. Και να τα πείτε αυτά και στο Συμβούλιο την επόμενη φορά που θα συζητηθεί το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όπως είπατε, αυτά που αποδίδει για τις δημόσιες επενδύσεις, για την ανακατεύθυνση οικονομίας. Αυτά είναι σωστά και τα παρακολουθήσαμε προσεκτικά. Δύο παρατηρήσεις λοιπόν που με ικανοποιούν. Η τρίτη τώρα έχει σχέση όταν είπα ότι θα πρέπει να είμαστε ή μηδέν αναστολή ή όχι αναστολή. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στα δύο. Μπορείτε να το σχολιάσετε. Αν δηλαδή δεν ε, ε, εκπληρώσετε τα πάντα, τότε μπλα μπλα μπλα μπλα. Ε, τότε, δηλαδή ή όχι αναστολή ή μηδέν αναστολή. Αναστολή με ένα αλλά μηδενική. Εγώ τα είπα αυτά και στους επιτρόπους. Εάν είστε ισχυρός και αρχίσετε τη συζήτηση με την Κομισιόν για ένα νέο όργανο, το οποίο θα ψηφίσουμε τότε το, το, το μήνα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτα στην Επιτροπή μας των Οικονομικών και μετά στην Περιφερειακή το νέο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και μπορείτε να ζητήσετε έξτρα υποστήριξη για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτά που είπε και ο συναδελφός μου πριν, ο κύριος Μπάλτς. Ίσως λοιπόν είναι σωστό ε, να σας δώσω τη συμβουλή να προσπαθείτε να το αρπάξετε αυτό το άλογο και να ανεβείτε πάνω. Ευχαριστώ κύριε Βανίστερο, κύριος Κοτσολίνο. Απαντήσατε κατά μεγάλο μέρος στις ερωτήσεις που θα σας έθετα για τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής εφόσον υπάρξει αναστολή και ακόμα και μόνο για το γεγονός ότι συζητήσαμε και συζητάμε εδώ και μήνες για την αναστολή. Τι αντίκτυπο μπορεί να έχει από την άποψη των ε, ε, δράσεων που πρέπει να λάβετε, τα μέτρα που προβλέπονται και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τη σχέση των ε, πολιτών με τα θεσμικά οργανικά της Πορτογαλίας και της Ευρώπης. Μας δώσατε λοιπόν απαντήσεις που με είναι ιδιαίτερως αλλά θα ήθελα να πω σε όλους Πραγματικά ίσως ε, φτάνουμε και προς το τέλος αυτής της συζήτησης, αλλά ήταν πολύ σημαντικός αυτός ο διαρθρωμένος διάλογος που έχουμε οργανώσει μεταξύ μόνη της Επιτροπής και με την ε, συμμετοχή των ε, Υπουργών της Ισπανίας και Πορτογαλίας. Θα πρέπει όμως να προσθέσουμε το εξής. Είναι μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και αυτό θα μπορούσε να σας ικανοποιεί και εσά στην Πορτογαλία και την Ισπανία, μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι ακόμη και η, όλη η ιδέα τη αναστολή των διευθυντικών ε, κομιτελίων, που για την Πορτογαλία έχουν μια άλλη ιδιαίτερη σημασία, είναι θέμα που πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Πρέπει να το ξαναμελετήσουμε και να προβλεφθεί διαφορετική νομοθεσία από ό,τι έχουμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε λάβει διαφορετικές θέσεις μεταξύ μας και μπορούμε να ξαναρχίσουμε μια συζήτηση σε άλλη φάση για ένα θέμα που ήδη συζητηθεί πολύ. Αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την πολιτική συνοχή ω ε, τιμωρητικό εργαλείο για να επιβάλλουμε τη μακρονομική πολιτική μα. Πραγματικά αυτό πρέπει να το ξαναδούμε και σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Λούερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Υπουργό. 27%, 27,2% βγάζει την ανεργία η Ευρωστάτη στην Πορτογαλία. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η ίδια με αυτή που έθεσα και στον κύριο Τεγκίνητος προηγουμένω, όπου δεν απάντησε. Ελπίζω να λάβω πορτογαλική απάντηση στην ερώτησή μου. Μπορείτε να μου δώσετε παραδείγματα πρωτοβουλειών, προγραμμάτων πρωτοβουλίας δηλαδή για την απασχόληση των νέων που δεν αποδίδουν και που θα έπρεπε είτε να επανεξεταστούν είτε να καταργηθούν και να ανακατευθυνθούν τα κονδύλια σε άλλα προγράμματα που θεωρείτε εσείς ότι μπορούν να αποδώσουν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βαν Μίλτενμπορκ των Φιλελευθέρων, Άλντε. Ευχαριστώ. Βεβαίω, η εφαρμογή του άρθρου 23 των κοινών διατάξεων είναι νομική υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ακούσαμε και από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριο Κατάινε. Δύο ερωτήσεις κύριε Υπουργέ συμφωνείτε ότι το κράτος δικαίου εφαρμόζεται και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στην Πορτογαλία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του άρθρου 23. Και δεύτερη ερώτηση, ποιες είναι οι δράσεις που έχουν αναλυφθεί ως τώρα και σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προετοιμαστεί η ενδεχόμενη αναστολή μέρους των πληρωμών των διαρθρωτικών ταμείων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κύριε Ομαρζή, Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Στα πλαίσια του διαθετικού διαλόγου είχα την ευκαιρία να πω ότι η ενδεχόμενη αυτή απόφαση για την αναστολή των πληρωμών των ταμείων είναι παράλογη, είναι επικίνδυνη και ε, καταλήγει τα αντίθετα αποτελέσματα. Και παράλογη, ειδικώ για την Πορτογαλία, που η Πορτογαλία σήμερα έχει λιγότερο σημαντικό έλλειμμα. Ε, το λιγότερο σημαντικό έλλειμμα εδώ και πολλές δεκαετίες. Επίσης είναι και ακατανόητη η απόφαση αυτή. Το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν βρήκε επαρκείς λόγους για να επιβάλλει χρηματικά πρόστιμα. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να βρει επιχειρημάτα, λόγους που να οδηγούν στην αναστολή των πληρωμών των ταμείων. Και να μην λησμονούμε το άρθρο 23. Το άρθρο 23 μίλει για ισότιμη μεταχείριση. Γιατί λοιπόν η Πορτογαλία γίνεται στόχος, γιατί όχι η Γαλλία, γιατί όχι η Γερμανία, σε ό,τι αφορά το ή τα πλεονάσματα της. Αυτές οι ερωτήσεις τίθενται. Δεν θα επανέλθω στα όσα ήδη λέχθηκαν, αλλά η ερώτηση που οφείλουμε να θέσουμε σε αυτούς είναι γιατί αυτό το παράλογο και αυτή η αυτό το ακατανόητο. μέσω αυτής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας να προσπαθήσουν να περάσουν δηλαδή μια σειρά διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων πολύ δύσπεπτων και κάποια στιγμή θα πρέπει η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον να θέσει ένα τέρμα στις προσπάθειες αυτές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάνα. Ευχαριστώ πολύ Βάνερ δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που προσήλθατε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, ευχαριστώ που τονίσατε και το σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι όντως αναγκαίο να γνωριζόμαστε και προσωπικά μέσα σε αυτόν τον διαρθρωτικό διάλογο. Επίσης είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο διαρθρωτικός διάλογος δεν τελειώνει σήμερα. Ότι θα πρέπει να τον συνεχίσουμε και άρα να επανέλθουμε και στη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τη ζητήσουμε να καταργήσει αυτό το παράλογο άρθρο 23 από τον κανονισμό των διαθετικών ταμείων. Έχω μια ερώτηση, την οποία έφυξε ακροθυγός μια προηγούμενη ομιλήτρια. Θέλω εγώ να εμβαθύνω λίγο. Ακούσαμε ότι ιδίω στην Πορτογαλία ήδη η απειλή της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας έχει οδηγήσει, έχει οδηγήσει, λέγω, στην αποφυγή λήψος επενδυτικών αποφάσεων και ιδίω έχουν παγώσει επενδύσει που επρόκειτο να γίνουν και με συγχρηματοδότηση από το Κοινωνικό Ταμείο. Μπορείτε να μα πείτε πιο συγκεκριμένα για ποια προγράμματα πρόκειται. Αν πρόκειται για προγράμματα για την καταπολέμηση τη φτώχεια ή τη ανεργία των νέων. καθώ επίση και ποιο είναι το εύρο των περικοπών. Είπατε επίση ότι τα διορθωτικά ταμεία είναι πολύ σημαντικά για δημόσιε και ιδιωτικέ επενδύσει στην Πορτογαλία. Βεβαίω εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σα και η έκθεση εκτελεστότητας λέει ότι οι επενδύσεις αυτές είναι μοναδικές για ορισμένες περιφέρειες. Μπορείτε να μας πείτε ποιες περιφέρειες θα πληγούν από τέτοιες περικοπές. Ευχαριστώ. μάθω, ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Υπουργέ που είστε εδώ. Το κίνημα των πεντεστέρων είναι κατά της μικροοικονομικής ερεσιμότητας είναι περιφέρειες που κι εσείς ο ίδιος στην επιστολή που αναφέρατε του Σεπτεμβρίου ε, θα επηρεαστούν ιδιαιτέρως. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο μια χώρα όπως η δική σας υποχρεώθηκε και επαναλαμβάνω υποχρεώθηκε να υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις ε, όπως αυτές που υλοποιήθηκαν πρέπει να τιμωρηθεί για το εργαλείο που βρίσκεται πιο κοντά στη ζωή των πολιτών. Το πλαίσιο αυτό δυσχεραίνει τη δουλειά της κυβέρνησής σας και προκειμένου να διασφαλίσει μια σχετική πρόοδο και να υπάρχει απαραίτητη κάλυψη στα πλαίσια της κοινωνικής προστασίας, ιδιαιτέρως με συστήματα εξασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος. Στις 6 Οκτωβρίου τρέχοντος ακούσαμε στην παρέμβαση της Επιτροπής ότι υπάρχει περίπτωση να ανασταλούν τα κονδύλια για το 2017. Πώ θα μπορέσετε να σχεδιάσετε με ασφάλεια το μέλλον σα, αν υπάρχει αυτή η πάθη να επικρέμεται από πάνω σα. Πώ μπορεί η πρόταση τη ε, ενισχυμένη πλειοψηφία να είναι κάτι που να το σκέφτονται σοβαρά στο Συμβούλιο. Είμαστε ενωμένοι εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο και θα πρέπει αυτά τα νομοθετικά κενά να τα ε, αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Συγγνώμη να σα διακόψω, ολοκληρώστε. Λοιπόν, επειδή έχουμε εντελώς ξεπεράσει το χρόνο, θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των άλλων επιτροπών για τη Δημοσιονομική Επιτροπή, ο κ. Φερνάντες, παρακαλώ. 1,5 λεπτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετώ τον Υπουργό και όλους τους συναδέλφους που είναι εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών Είμαστε κατά τη αναστολή των Ευρωπαϊκών Διευθυντικών Κονδυλίων και Επενδυτικών Κονδυλίων για την Πορτογαλία. Το έλλειμμα του 2015 έφτασε κάτω από το 3% με 98% μείωση βάσει της Εθνικής Στατιστικής μας Υπηρεσίας. Οπότε πρέπει να πάψει και η διαδικασία για το προβολικό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι η Πορτογαλία σεβάστηκε το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η διαδικασία για το υπερβολικό έλλειμμα δεν θα έπρεπε καν να έχει ξεκινήσει. Εδώ επίσης αληθεύει ότι ο διερθωμένος διάλογος θα πρέπει να οδηγήσει ώστε οι συζητήσεις μας αυτές, όπως δείχνει η συντριπτική πλειοψηφία, ε, θα πρέπει να εισακουστεί για την μη εφαρμογή ε, αυτής της απόφασης, της ενδεχόμενης απόφασης για την αναστολή των διευθυντικών κονδυλίων. Είδαμε πώ επιζήμια θα είναι αυτά τα μέτρα κατά τη οικονομία, κατά των νέων, κατά των αλλαίων, κατά των ε, ε, επιχειρηματιών. Πόσο θα υπονομευθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μία ερώτηση λοιπόν προ τον Υπουργό. Υπάρχει κάποια, ε, κάποιο στόχο, κάποια δέσμευση που έχει αναλάβει η κυβέρνηση φέτο για τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματο που έπρεπε να έχει εφαρμόσει και δεν έχει εφαρμοστεί. Και τι αντίδραση θα υπήρχε όπως, ως προς την υλοποίηση των ε, μέτρων που ήδη έχουν προβλεφθεί για την κάλυψη του ελλείμματος και την ανάπτυξη. Ευχαριστούμε κυρία Ριμπέρο από την Επιτροπή Επασχόλησης. Ευχαριστώ η Επιτροπή που α, εκπροσωπώ απέρριψε την επιβολή της αναστολής κατά της Πορτογαλίας και ήμουν εισηγήτρια για αυτό το σώμα. Θεωρούμε ότι η διαδικασία για το υπερβολικό έλλειμμα ε, προχώρησε χωρίς την απαραίτητη αιτιολόγηση. Με γραπτή μα ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τον Ιούνιο, εντοπίσαμε την τεράστια προσπάθεια των Πορτογάλων από το 2011, που οδήγησε σε σημαντική μείωση του ελλείμματο επί 4 χρόνια κατά 17% τουλάχιστον, και αυτό από μόνο του θα εξηγούσε το γιατί πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα και καμία ε, φυσικά ποινή ή αναστολή. Η όλη αυτή η συζήτηση τίχνεται θα, να, θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν η πορτογαλική κυβέρνηση είχε εξηγήσει, είχε μάλλον να θέσει ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, την, για τον όγκο του πορτογαλικού ελλείμματος που ήταν το 2015 δηλαδή κάτω από το 3% όπως ορίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Έχουμε όλες τις συνθήκες για να μπορέσουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό μια για πάντα. Όμω βλέπουμε να υπάρχουν μακεδελικέ προθέσει κατά τη Πορτογαλία, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι όλα αυτά τα θέματα δεν έχουν, ε, όπω η αναστολή δεν θα έχει καμία, κανένα κοινωνικό αντίκτυπο, διότι οι προσπάθειε για την ενίσχυση τι απασχόλησει και την καταπολέμηση τη φτώχεια από το 2009 έχουν ε, επιδιωθεί σωστά από την Πορτογαλική κυβέρνηση. Μα εδώ τη θέση αυτή την έχετε ακούσει και τη συμμερίζονται όλοι εδώ. Το Κοινοβούλιο αριστερά και δεξιά υπερασπίζεται ε, αυτή την γραμμή και στην Πορτογαλία υπάρχει και η ίδια ευθύνη. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε ότι να ακολουθήσουμε μία από τις δύο επιλογές. Ή ε, θα συνεχιστεί αυτή η γελία διαδικασία που ε, πραγματικά υπονομεύει την ίδια μας τη χώρα εις βάρος και των Πορτογάλων πολιτών και της ευρωπαϊκής προσπάθειας και βεβαίως των μελλοντικών προοπτικών ολόκληρης της χώρας. Ευχαριστούμε. Έχουμε εκπροσώπους από την Επιτροπή Άγκρη. Ευχαριστούμε ως Μέλου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Για μια φορά εδώ δεν ε, θα περίμενε κανείς να έχει υπουργό σοσιαλιστή και κάποιον εκπρόσωπο της αντιπολίτευσης για να συζητήσουν. Πρέπει να πω όμω ότι η διαδικασία αυτή είναι μια διαδικασία που ε, υπονομεύει την Ευρώπη και είναι για την Πορτογαλία. Εδώ, αν δούμε τι αποτέλεσμα είχαν τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο 2015, το έλλειμμα κατέβηκε από το 3%. Αυτό σημαίνει ότι η Πορτογαλία παρήγαγε ένα έλλειμμα ε, κάτω του 3%. Το πλεόνασμά μας ξεπέρασε δηλαδή ε, αυτό που οριζόταν ως στόχο και τώρα μπορεί να είμαστε θύματα ε, του να μας επιβληθούν κυρώσεις. Πρόσφατα το είπε και ο Επίτροπος Μοσχοβησή για τα θέματα αυτά και ο Επίτροπος το και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι κυρώσεις κατά της Πορτογαλίας θα πετύχουν στη χώρα το αντίθετο από αυτό που έχει απαιτηθεί ως τώρα. Α, ας δούμε δύο λεπτά. Ε, αυτό που είπε και ο Γάλλος πρόεδρος ε, προς στιγμήν, ε, ο Βαπάντιρ δεν θα το πούμε έτσι δηλαδή, αν ληφθεί μια τέτοια πρέπει, ε, απόφαση. Εδώ πρέπει να ενωθούν όλες οι δυνάμεις για να εμποδίσουμε αυτήν την απόφαση. Αυτό πάντως που θέλω να πω προς τον πρόεδρο Ολάντ είναι ότι εμείς από την Πορτογαλία όπως η Γαλλία έχουμε τις δικές μας ένοπλες δυνάμεις, έχουμε και διπλωματικές δυνάμεις και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ιστορία ούτε είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε για τις ένοπλες δυνάμεις και την άμυνα της Γαλλίας. Ε, Κύριε Υπουργέ και Πρόεδρε, η Γαλλία είναι η Γαλλία και τη σέβομαι απεριόριστα. Όμω και η Πορτογαλία είναι Πορτογαλία. Και πρέπει και αυτή να τη σεβαστούμε. Σα παρακαλώ, κύριε Μέλου. Σα παρακαλώ. Δεν είχα την ευκαιρία να δώσω το λόγο στου προσωπικού. Ε, εκπροσώπου. Από την. Ε, Ο κύριο Φερέιρα τώρα έχει το λόγο. Την επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το απλό γεγονός ότι βρίσκεται εδώ ο Υπουργός δείχνει ότι όλη η διαδικασία είναι απαράδεκτη. Πίεση εις βάρος της Πορτογαλίας, προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης, ε, προσπάθεια ε, ε, ομοιρίας του πορτογαλικού λαού. Ήδη αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε για τη ρήξη με τις πολιτικές που προσπαθεί να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιλάμε για την ενδεχόμενη αναστολή των διευθυντικών και επενδυτικών κονδυλίων προς την Πορτογαλία. Απαράδεκτη ήδη λογική, λόγω των όσων εκτέθηκαν και πολλών ακόμη. Θέλω όμως να πω το ακόλουθο τα διδοτικά κονδύλια που προβλέπονται για την Πορτογαλία από το 14 έως το 20 ξεπερνούν κατά λίγο τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επενδυτικά κονδύλια είτε για την Πορτογαλία είτε για την ανακόφηση του χρέους ε, ε, είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. Το διπλάσιο από τα ε, διαστατικά και επενδυτικά κονδύλια που προβλέπονται. Οι ευθύνε λοιπόν των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων που συνεχίζουν να εθελοτυφλούν είναι τεράστιε. Δεν υπάρχει καμία συνοχή και δεν μπορούμε να αγνοούμε την ε, πίεση αυτή που επιβάλλεται στην Πορτογαλία, την πίεση αυτή με το χρέο και το πόσο χρειάζεται επενδύσει η χώρα αυτή για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση για να εξορροπηθούν και πάλι οι λογαριασμοί και οι πληρωμέ τα διάφορα στοιχεία του προπολογισμού. Εάν συνεχίσουμε έτσι, θα προλάβουμε να ακούσουμε τον Υπουργό στο τέλο τη συνεδρίαση. Δύο ακόμα εκπροσώπου τη Επιτροπή Ρέτζη, ο κύριο Ζούρε και η κυρία Ροντρίγκε. Σα παρακαλώ, μπορείτε σε τρία δευτερόλεπτα να μα πείτε αυτό που θέλετε να πείτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με όσοι υπόθηκαν εδώ δεν είναι εύκολο να καταλήξουμε σε μια. Μάλλον δεν είναι δύσκολο να ολοκληρώσει κανεί και να καταλήξει ένα λογικό συμπέρασμα. Η κεντρική κυβέρνηση δεν μπορεί να ε, τιμωρηθεί και έτσι να υποβληθούν τόσες, ε, να επιβληθεί αυτή η τιμωρία σε ολόκληρη τη χώρα. Βλέπουμε ότι με τους λογαριασμούς μας και τον προπολογισμό φτάσαμε περίπου τους στόχους που προβλέπονταν. και με την ε, αναθεώρηση, με τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, καταφέραμε πολύ περισσότερα ε, και ως Πορτογαλία, αλλά το ίδιο και στην Ισπανία. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, χρειάζονται κανόνες. Και οι κανόνες, ε, εφόσον τηρούνται, θα πρέπει να υπάρχει μια ευελιξία. Θα κλείσω, Πρόεδρε. Ε, πρέπει να σας διακόψω. Πρέπει να σας διακόψω, διότι δεν μπορούμε να ακούσουμε, δεν ακούσουμε τον Υπουργό έτσι. Κύριε Ροντρίγκε, 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ γρήγορη. Εδώ είναι προφανές ότι προσπαθούμε να διακόψουμε, να υπάρξει ρήξη με την παράλογη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Κύριε Υπουργέ, μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς βλέπετε την ενδεχόμενη αναστολή των κονδυλίων, όπως προβλέπουν οι συνθήκες λένε ότι είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την διόρθωση των μικροοικονομικών ανισορροπιών στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχετε το λόγο. Ο χρόνος μας είναι λίγος. Ελπίζω να μπορέσετε να απαντήσετε τα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και θα συνδυάσω διαφορετικά θέματα, προσπαθώντας να αποφύγω σε κάθε έναν ξεχωριστά και θα μιλήσω αγγλικά. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε στα πορτογαλικά. Αυτό που θέλω να πω, απαντώντας σε ένα θέμα που έθιξαν πολλοί από τους ε, βουλευτές, είναι ότι η αναστολή των ε, κονδυλίων πρέπει να ε, ακυρωθεί με όλη τη σαφήνεια που πρέπει. Είναι απαραίτητη η σαφής ακύρωση. Πρέπει να προβληθούν σωστά οι στόχοι που επιδιώκουμε και να γίνουν κατανοητοί και από τον ε, πληθυσμό, από τους πολίτες τους πολίτες αυτούς για τους οποίους εφαρμόζουμε τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό έχουμε το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Γι' αυτό έχουμε μια πολιτική πραγματικά συνεκτική. Αυτήν την ε, πολιτική συνοχής που επιζητά και την ανάπτυξη. Την ανάπτυξη όπου θέλουμε όλοι να έχουν συμμετοχή. Μια ε, επένδυση που θα προσελκύσει περισσότερο κόσμο στην αγορά εργασίας είδαμε πόσο με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Πορτογαλία χάσαμε τόσους νέους νέους που αυτοί είναι ουσιαστικά οι δικαιούχοι, αυτοί στους οποίους απευθύνεται η πολιτική συνοχή. Η ενδεχόμενη αναστολή λοιπόν των κονδυλίων τέτοιου είδους κινήσεις είναι αποφάσεις που πλήττουν την απασχόληση των νέων. Ε, αξιολογούμε διαρκώς τις ε, ενεργές πολιτικές που αφορούν ακριβώς αυτή την ηλικιακή ομάδα. Η μεταβολή των δημογραφικών τάσεων ή των μεταναστευτικών τάσεων ή της οικονομικής ανάπτυξης μπορεί ακριβώς να μας επιτρέψουν να επενδύσουμε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα και θα ε, πληγούν όλος ιδιαίτερος από μια οποιαδήποτε αλλαγή στα διαδικτικά κονδύλια. Οι περιοχές, οι γεωγραφικές περιοχές που θα επλήττουν το περισσότερο από την ενδεχόμενη αναστολή είναι προφανώς οι περιοχές της ΥΠΕΔ, του εσωτερικού της χώρας. Είναι περιοχές όπου κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος των κοινοτικών κονδυλίων και η διάσταση της εδαφικής συνοχής που είναι πολύ σημαντική για τη χώρα, ιδίως με το Εθνικό Πρόγραμμα των Μεταρρυθμίσεων, που είναι ένας από τους πυλώνες της εδαφικής ε, συνοχής, είναι κάτι που προασπίστηκε με ιδιαίτερη θέρμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κονδύλια λοιπόν είναι άκρο σημαντικά για αυτήν τη διάσταση. Βεβαίω, δεν έχουμε σενάρια για το ποια θα ήταν τα έργα που θα κυρώνονταν, διότι έχουμε εμπιστοσύνη ότι έχουμε κάνει ό,τι πρέπει και ότι έχουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα για να μην υπάρξει αναστολή. Τα μέτρα που ευαγγελιζόμαστε για την ανάπτυξη της Ευρώπης είναι μέτρα που από την πολιτική τους φύση στόχο έχουν να κάνουν την Ευρώπη να μην είναι απλώς ε, ένας τόμος ε, γεμάτος από κανόνες. Θέλουμε μια Ευρώπη για τους πολίτες. Και αυτή την Ευρώπη οι πολίτες πρέπει να την καταλαβαίνουν και να την ακούν. Δεν υπάρχει λόγος για την αναστολή των κονδυλίων με μια οικονομία που σέβεται τους στόχους της. Με μια οικονομία που στην πάρα των ετών έχει ακολουθήσει τόσο προβλέπουν οι συνθήκες και η ευρωπαϊκή της ε, πορεία. Θα συνεχίσουμε να εμένουμε προς αυτή την κατεύθυνση και αν υπάρχουν ως προς αυτό αμφισβητήσεις, δυστυχώς υπονομεύεται η εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή, στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Υπονομεύεται ίδια της η συνοχή. Γι' αυτό και πιστεύουμε και επιμένουμε ότι αυτός ο μηχανισμός δεν είναι αποτελεσματικός για την πρόθεση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης. δεν συμπαρασύρει τους πολίτες προς το στόχο του εγχειρήματο. Και η όλη συζήτηση των κονδυλίων πλήττει τομείς εξαιρετικά ευαίσθητους που μιλάμε εδώ για χώρες οι οποίες έχουν πλήρη συνείδηση, ε, θέλουν να κάνουν κάθε βήμα που χρειάζεται για να προχωρήσουν, όλα έχουν λάβει σάρκα και οστά και σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση που τοποθετούμεθα. Θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Πορτογαλία τηρεί μια στάση ιδιαίτερα θετική, είναι θετικά διακείμενη προς την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό πνεύμα που διαπνέει τους ε, πολίτες της χώρας, το έθνος μας, πραγματικά φαίνεται από την αφοσίωση που έχουμε δείξει στην επίτευξη των στόχων μας και θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία, μια πορεία που θα φέρει ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ελπίζουμε ότι θα φέρει ανάπτυξη στην κάθε μια γεωγραφική περιοχή ξεχωριστά και το κάθε ευρωπαϊκό έθνος. Είναι μια, μια υπόσχεση που έλαβε η, Ευρωπαϊ... η Πορτογαλία από τότε που προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση και είναι και μία δέσμευση που έχουν αναλάβει όλες οι πορτογαλικές κυβερνήσεις ως σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύρια, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ όλες τις λεπτομερεί ε, ευχαριστώ για τις λεπτομερείς απαντήσεις μάλλον, ελπίζω να απαντήσατε στα ερωτήματα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Γκουαλτιέρη για να κλείσει τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ όπως υπογράμμισε ο κ. Βανίστελρο, ήταν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και χρήσιμη διαδικασία διαλόγου και νομίζω ότι είμαστε όλοι αισιόδοξοι ανεξάρτητα από το πώς βλέπουμε μακροοικονομικά ε, το μακροοικονομικό αυτό εργαλείο, έχουμε ποια είναι η θέση μας, ε, για να μην υποβάλει η Κομισιόν ε, κανένα, ε, καμιά πρόταση αναστολής, χρειάζεται κάποιες προϋποθέσεις και νομίζω ότι πληρώνουν εδώ ε, και συνεισφέρουμε και εμείς ε, για να αποφευχθούν έτσι παράλογες, ε, μη ορθολογικές συμπεριφορές και μη κατανοητές. Ήταν νομίζω χρήσιμη, χρήσιμος διάλογος, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό, αλλά θα πρέπει πρώτα να αξιολογήσουμε, να το αξιολογήσουμε αυτό, να, να μείνουν συντονιστές λίγα λεπτά. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ και τις διερμηνείς ε, ο κ. Γουαλτιέρη για τις προσπαθίες τους.